Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να αρχίσουμε, εάν θέλετε, με το πρώτο σημείο της ημερησίας ε, διατάξεως, δηλαδή την έγκριση της ίδιας και βέβαια έχουμε και το γλωσσικό καθεστώς με τις εξής γλώσσες. Θα σας πω τις γλώσσες που δεν θα μεταφράζονται βουλγαρικά, δανέζικα, εστονικά, φιλανδικά, ουγγρικά, κελτικά, ιρλανδικά δηλαδή και ορισμένα άλλα μεταξύ αυτών πορτογαλικά, πάντως τα ελληνικά μεταφράζονται. Και αυτό συμβαίνει διότι, συνεχίζει ο πρόεδρος, έχουν προτεραιότητα για ύπαρξη μεταφραστών μόνο οι γλώσσες των τακτικών μελών. Οι μητρικές γλώσσες δηλαδή των τακτικών μελών. Εάν δεν έχετε ενστάσεις, εγκρίνεται η ημερησία διάταξης. Και ας προχωρήσουμε αμέσως στο θέμα του υπαρθμόν 3 ε. την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη European Facility δηλαδή και έχουμε την κυρία Ράινες Τσοβανίδες και τον κύριο Τέρι Μουσέρ. Ε, θα αρχίσουμε την επί συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την πρόοδο της European Peace Facility. Την έχουμε βάλει αυτήν στην ημερήσια διάταξη από εδώ και δύο εβδομάδες ε, όπου το Συμβούλιο Υπουργών εξέφρασε επιφυλάξεις για το πεδίο εφαρμογή της EPF και ζήτησε να γίνει περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου και θα θέλαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατανοήσουμε κατά πόσο μπορεί να επανεξεταστεί το υφιστάμενο πλαίσιο. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Βάουτμανς. Ε, δυστυχώς δεν την βλέπω να είναι παρούσα ακόμη. Η κυρία Βάουτμανς συμφώνησε να αναβληθεί η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2019. Και παρακαλεί να ληφθούν υπόψη από τους συναδέλφους οι σημερινές συζητήσεις καθώς και ανταλλαγές απόψεων με την ύπατη εκπρόσωπο όταν δηλαδή θα υποβάλουν τροπολογίες οι συνάδελφοι. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα θα διαβιβαστεί στους, στα μέλη από την γραμματεία μετά από την συνεδρίαση. Λοιπόν, ξαναλέω, Ας δώσουμε τον λόγο πρώτα στον κύριο Τιρί Μουσέρ, Policy Officer, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μουσέρ, EAS, μέλος μικρής ομάδας που συντάσσει και διαπραγματεύεται την European Peace Facility στο Συμβούλιο υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα Σερανό. Η European Peace Facility θα χρηματοδοτήσει τρεις δράσεις CFSP και πάντα δηλαδή, άμεσες επιχειρήσεις με μηχανισμό που ονομάζεται Αθήνα, μετά μέτρα capacity building για τις υποδομές των ενόπλων δυνάμεων των εταίρων μας και τέλος στήριξη ειρηνευτικών αποστολών τρίτων όπως η Αφρικανική Ένωση. Ο στόχος της EPF, European Peace Facility, είναι να ενισχύσει την ικανότητα να δρουν σε, στα πλαίσια ειρηνευτικών αποστολών αποκατάστασης ή διατήρησης και η ιδέα είναι ότι έως τώρα είχαμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε δράσεις στους τομείς αυτούς όπως για παράδειγμα η αποστολή στη Σομαλία και πιο πρόσφατα στη Σαχέλ, η Αφινά χρηματοδοτεί άμεσα επιχειρήσεις, σημειώνονται όμως κενά. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε δράσεις εκτός της Αφρικανικής Ένωσης. Διότι δεν είναι επιλέξιμα ορισμένα, δεν είναι επιλέξιμες ορισμένες δράσεις για χρηματοδότηση το γεγονός, για παράδειγμα, ότι όταν έχουμε νέα εκπαιδευτική αποστολή, το πρόβλημα είναι η μεταφορά των κληρωτών εκεί όπου θα εκπαιδευτούν, καθώς και μεταφορά εξοπλισμού. Και μεταφορά τους πάλι προς τα πίσω ή μάλλον εκεί όπου θα ε, δραστηριοποιηθούν επιχειρησιακά. Αυτό λείπει για την ώρα. Η Αφίνα δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει αυτά γιατί δεν εντάσσονται σε αποστολές ΝΑΤΟ. Η EPF λοιπόν δεν θα έχει όρια σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες χρηματοδοτήσεις, ούτε γεωγραφικές. Θα υπάρχουν βέβαια περιορισμοί σε ό,τι αφορά την δράση που θα αναλαμβάνει, αλλά αυτό θα κρίνεται αναπερίπτωση, όταν δηλαδή θα εγκρίνεται η κάθε συγκεκριμένη δράση. Αρχίσαμε από τα μέσα Ιουνίου με παρουσιάσεις στην Κορεπέρ και στις άλλες συναρμόδιες ομάδες, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Προχωρήσαμε στις διαπραγματεύσεις στην ομάδα η οποία αναλαμβάνει ε, τις να προχωθεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και για την ώρα συζητούμε τους λόγους για τους οποίους η European Peace Facility έχει προταθεί και με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Συζητούμε δηλαδή τα γύρω-γύρω από την EPF και όχι την ίδια την EPF. Θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το κείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου τον Ιανουάριο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που διαθέτουμε και αναμένουμε βέβαια μακρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για κάθε ένα άρθρο ξεχωριστά καθώς και για το εάν θα υπάρξουν τροπολογίε που ρώτησε ο Πρόεδρος, βεβαίω θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες για το κείμενο. Το αναμένουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Εσείς κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Συνδέσμου της EPF για συνεργασία με οργανώσεις ανά τον κόσμο, για την πρόληψη συγκρούσεων. Έχουμε μακρότατη εμπειρία σε, στα πλαίσια συγκρούσεων και για την προστασία τοπικών κοινωνιών, αλλά και σε επίπεδο κρατικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ανάμεσα σε αυτό και στα Εθνικά Κοινοβούλια και αρχίζουμε να εξετάζουμε την EPF Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για την αφετηρία μια διαδικασία συζητήσεων. Η παρέμβασή μου λοιπόν μάλλον θα θέσει περισσότερα ερωτήματα παρά να δώσει απαντήσεις. Θέλω να τονίσω ότι η προτινόμενη Peace Facility αποτελεί απόκληση από τις συνήθει δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το ιστορικό της που είναι ότι προωθεί την ειρήνη, δηλαδή δεν πρόκειται για business as usual. Προτείνεται μια ε, διαδικασία διευκόλυνσης της Ευρώπης για την χορήγηση ε, πολεμεφοδίων καθώς και των ε, μισθολογίων των ε, στρατιωτικών με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Λαμβάνουμε λοιπόν μια διαφορετική κατεύθυνση. Τρία αφηγήματα στρέφονται γύρω από την πρόταση. Το ένα είναι ότι κάθε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην ειρήνη και δεν κάνει κακό. Δεύτερο, ότι φέρει την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει αυτόν τον προωθητικό ρόλο. Επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που το κάνει δεν μπορεί να κάνει κακό. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να αμφισβητηθεί. Ένα άλλο αφήγημα που κυκλοφορεί είναι γύρω από την πρόταση, το επιχείρημα δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το δύσκολο και προκλητικό περιβάλλον χρειάζεται να έχει και hard power και όχι μόνο soft power για να δράσει παγκόσμια. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται ε, να αποστασιοποιηθούμε κάπως. Είναι σαφές ότι η πρόταση φύγει μια ευαίσθητη χορδή της δράσης της Ένωσης, αλλά ας εξετάσουμε τα μέτρα εκπαίδευσης και εξοπλισμού τα οποία υλοποιούνται από άλλες χώρες στην Συρία, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και τότε θα δούμε πώς αποδίδουν αυτά τα μέτρα. Άλλο αφήγημα πάλι γύρω από την ίδια πρόταση είναι ότι ενδεχομένως αποτελεί λύση απέναντι στον εξτρεμισμό που αισθάνονται πολλές χώρες αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δούμε και αυτό το πράγμα με κάποια απόσταση, θα δούμε ότι όλο και περισσότερε οργανώσει και οντότητε διεξάγουν έρευνε για τι αιτίε που οδηγούν ε, διαφόρου να συμμετάσχουν σε τέτοιε ομάδε και αυτό είναι και η βία αντιμετώπιση του από τις δυνάμεις Ε, Αν δείτε και κάποιε προτώσεις που γίνονται, αυτέ προκαλούν ανησυχία, διότι ο κόσμο φοβάται για την ασφάλεια τη διατροφή, για παράδειγμα. Πρέπει και εδώ λοιπόν να αποστασιοποιηθούμε λίγο από αυτό το αφήγημα. Επαναλαμβάνω ότι ωστόσο δεν πρόκειται για business as usual και πρέπει να εξεταστεί με κριτικό πνεύμα. Το σχέδιο εκθέσεως της κυρίας Χόμπατμαν μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλά από τα πράγματα αυτά και κυρίως ότι χρειάζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος που δεν υφίσταται για την ώρα. Θα ε, υποστηρίξουμε λοιπόν πολύ το επιχείρημα που περιλαμβάνει στο σχέδιο εκθέσεώς της εισηγήτρια σχετικά με την θέσπιση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ. Τώρα, για την λίστα των ερωτήσεων, πρέπει να δούμε πώς η προτινόμενη European Peace Facility θα ενισχύσει την ανθρώπινη ασφάλεια. Θα χρειαστεί να εξηγηθεί αυτό περισσότερο στην πρόταση. Πώς θα προωθήσει την ανθρώπινη ασφάλεια. Ο τίτλος του προτινόμενου μηχανισμού είναι παραπλανητικός, διότι δεν υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση. Τι είδους ανάλυση κινδύνου θα πρέπει να γίνει ώστε, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επέλθει κίνδυνος, ότι θα μετριαστούν τα δεινά που ενδεχομένω υφίστανται οι άνθρωποι κλπ επειδή υπάρχουν και σημαντικά επίπεδα διαφθοράς και βεβαίως και μέσα στον παγκόσμιο ανταγωνιστικό εμπόριο εξοπλισμών, τι μέτρα θα ληφθούν και μηχανισμοί θα θεσπιστούν ώστε η European Peace Facility να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση που θα δίνει θα χρησιμοποιείται σωστά. Επίσης, η συνοχή των δράσεων της European Peace Facility πώς θα εξασφαλιστεί όταν μιλούμε για συνοχή πώς θα συνέχεται με άλλες εξωτερικές δράσεις, μέτρα διατήρησης της αρήνης, του άρθρου 28, ε, sector reform, καθώς και άλλες δράσεις που αναλαμβάνουν, αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Υπάρχει και η African Peace Facility και εκεί έχει αυτή η μηχανισμό λήψης αποφάσεων, αλλά το αφήνουμε αυτό για την ώρα. Πρέπει να δούμε εάν πρόκειται για έναν τρόπο με τον οποίο οι χώρες μέλη μπορούν να παρέχουν εξοπλισμό σε χώρες εταίρους με τρόπο που τα κοινοβούλια τους δεν θα δέχονταν. Ενώ λοιπόν ίσως να υποστηρίζεται από τους πολιτικούς αυτή η, αυτής η δράση εξοπλισμού, όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται, μπορεί να μην την υποστηρίξουν την πρόταση. Πάλι μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην δημιουργία ικανότητας, capacity building δηλαδή, και στην ευρεία δράση για την εξασφάλιση της ειρήνης, αλλά είναι δύσκολο να βρεθούν ε, project τα οποία θα χρηματοδοτηθούν. Μας έχουν πει ότι λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, διότι αυτό βρίσκεται μέσα στο DNA της Ευρώπης. Αλλά μέχρι τώρα κανένας δεν μας έχει εξηγήσει πώς θα εξασφαλιστεί αυτό στην πράξη εγώ δεν κατανοώ ποια είναι η προστιθέμενη αξία για την παροχή υποστήριξης, εκπαίδευσης και εξοπλισμού σε χώρες εταίρους υπό τον Ευρωπαϊκό Αυτομηχανισμό. Ποιο είναι το πλεονέκτημα που προσφέρει και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουρες ότι οι κίνδυνοι μετρούνται επαρκώς και επιπροσθέτως. Αυτοί που θα επιβλέπουν τον μηχανισμό έχουν σχετική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ε, αποκατάσταση της ειρήνης για τον να γνωρίζουν πού πηγαίνουν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις. Πάλι για το CBST που περιλαμβάνεται στην πρόταση και στον μηχανισμό και εκεί προστίθεται ο νέος αυτός μηχανισμός, πώς όλα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους και πρόκειται για υψηλή χρηματοδότηση. Όπω είπα λοιπόν στην αρχή τη ομιλία μου, πρόκειται για την αφετηρία μια συζητήσεω. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα επιμέρου στοιχεία από την πλευρά τη κοινωνία των πολιτών, με τη βοήθεια οργανώσεων οι οποίε ε, εργάζονται από δεκαετιών για το θέμα αυτό. Και ε, για την ώρα δηλώνω ότι δεν είμαι ικανοποιημένη από τι προφορίε που παρέχονται. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα λοιπόν ε, πρέπει να οργανώσουμε κάπως τη συζήτηση. Προτείνω να ξεκινήσουμε με την κυρία Οτμάν. Then, ε, shadow reporters, Mr. Μετά τους κύριο του κύριο Γκάντζαν. Κύριε Σπίτσουλα, θέλετε. και μετά μπορούν να απαντήσουν και οι δύο προσκεκλημένοι μας όποιες ερωτήσεις υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε ε, ευχαριστώ κύριε, κύριε Κοιτάξτε, έχω μείνει έκπληκτος από αυτά που ακούω. Αγαπητή κυρία, ο οργανισμός σας δεν είναι ο μόνος με επαγγελματίε που γνωρίζουν τι σειράξει, ε, τι επιλύσει των κρίσεων, τη διαχείριση των προγραμμάτων ασφαλεία. Υπάρχει κόσμο ε, στην Κομισιόν, εδώ στο Κοινοβούλιο, στι στρατιωτικέ μα δυνάμει. Ε, δεν είναι βρισιά οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας με αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα ασφαλεία, προγράμματα μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας το μονοπόλιο λοιπόν που θεωρείτε πρέπει να έχετε για να βαθμολογήσετε θετικά και αρνητικά αυτή την πρόταση μου φαίνεται τρομακτικό θράσος. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τίποτα δεν είναι γραμμένο πουθενά το οποίο να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικαστεί στο να μην έχει ποτέ hard security και να μην ασχοληθεί με στρατιωτικά ζητήματα. Υπάρχει η ΠΕΣΤΕ, υπάρχουν στρατιωτικέ ε, δράσει και επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην αρέσουν σε πολλού, αλλά υπάρχουν. Σε μέτριο βαθμό φυσικά. Προβλέπουμε και ένα εργαλείο το οποίο θα κάνει κάποια πράγματα παραπάνω στο στρατιωτικό τομέα. Ε, και να γίνουμε ξαφνικά, λέτε εσεί, σε μια στρατιωτικοποιημένη οργάνωση και να κάνουμε μόνο αυτό. Λοιπόν, από μία είναι εύλογο να κάνουμε ερωτήσεις ε, και εκτενείς ε, και εγώ ήμουν ε, για το μηχανισμό CBSD εισηγητής. Να σας πω ότι το πήγαμε στο ελάχιστο, στο ό,τι πιο ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε σε θέματα ασφαλείας για να λάβουμε υπόψη τα οικονομικά, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πάντα. Είναι λοιπόν λογικό που κάνουμε τη συζήτηση εκεί τώρα για την πλαισίωση, για τον έλεγχο αλλά σε τελική ανάλυση γιατί συστηματικά τέτοιες προθέσεις για θέματα στρατιωτικής ασφάλειας. Τέτοια δίκη προθέσεων. Εγώ θέλω να μην, προτιμώ να μην ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ζήτημα καθόλου, αλλά οι άλλοι θα ασχοληθούν και όλες οι ερωτήσεις που κάνετε σήμερα στους Ευρωπαίους πηγαίνετε να τις κάνετε Στου Τούρκου, στους ρώσου, στους Κινέζους για να δείτε πώς ασχολούνται αυτοί με τη λογιστική, με τη διαφθορά, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τις κοινοβουλευτικέ ευθύνε. Γιατί είναι ωραία να λέμε ότι εμείς είμαστε οι κακοί της διεθνού κοινότητας διότι θέλουμε να επενδύσουμε λίγο παραπάνω σε αυτά τα ζητήματα τη ασφάλεια. Αλλά εξηγήστε μου, αν θέλετε, τι θα κάνουμε. Αν δεν έχουμε τα μέσα να Έχουμε κάποια πράγματα και το κάνουν άλλοι. Πάρτε για παράδειγμα την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ένα κράτο τελείω κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν υποδομέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά και στηρίζει, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες. Ειδικότερα στα προγράμματα εκπαίδευση και εξοπλισμού, τα train and equip, όλα αυτά που φαίνεται να δαιμονοποιούνται από διάφορους. Ποιο θα κάνει το train and equip λοιπόν εκεί, οι Ρώσοι. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερη λύση. Θεωρείτε ότι αυτοί θα σέβονται καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο για την κεντροαφρικανική δημοκρατία να ασχοληθεί μαζί τη η Ρωσία αντί για εμά. Εγώ θεωρώ όχι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συνέχεια στι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια συνέχεια από τη στιγμή που εμπλέκεται διπλωματικά, ε, ενδεχομένω και στρατιωτικά με τις αναπτυξιακές πολιτικές που είναι πολύ στιβαρές και τις οποίες υλοποιεί και μετά κατά καιρού ε, υπάρχει και κάποια ανάγκη σε θέματα ασφάλειας, στήριξης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, train and equip. Α μην γελιοποιούμε λοιπόν τη συζήτηση, γιατί αυτό που άκουσα τώρα ήταν γελιοποίηση τη συζήτηση. Ναι, τίθενται διάφορα ερωτήματα και εμεί πρέπει να θέσουμε διάφορα ερωτήματα ω ε, βουλευτέ ε, για τον έλεγχο, την οργάνωση, τη διακυβέρνηση αυτού του εργαλείου. Αλλά σα συγκετεύω, μην μα ξεκινάτε αυτή την αστεία ε, αμφισβήτηση κάθε φορά που πάει να ασχοληθεί με κάτι στρατιωτικό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κακό, είναι βρώμικο και σίγουρα μεροληπτικό. Εντάξει, μπορούμε να ασχοληθούμε για να είναι κάπως καλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά το να μου λέτε ότι στρατιωτικοποιούμε υπερβολικά τα εργαλεία μας και ότι οδηγούμαστε σε καταστρεπτικά αποτελέσματα είναι υπερβολή. Ας σταματήσουμε λοιπόν όλο αυτό τον τρόπο, όλο αυτό το διήγημα που συνοδεύει αυτό το οικονομικό εργαλείο και το αντεπιχείρημα όπου κάθε προσπάθεια να εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο αμυντικό εργαλείο λέμε ότι διαστρεβλώνει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριο Γιούρεκ ε, δεν επιθυμεί να ομιλήσει ο κύριος Γιούρεκ και επανερχόμαστε λοιπόν σε εσά, ε, κυρία. Μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Μπουσέρ. Ορίστε εσείς πρώτοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα τη μετάφραση, ελπίζω λοιπόν να μην έχασα τίποτα. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω τα σχόλιά σα, αλλά κάπως Παραφράσατε τα όσα είπα. Ε, δεν επηρεάζομαι ούτε από τους Ρώσους ούτε από τους Κινέζους. Δεν είπα αυτά τα πράγματα. Βρίσκομαι εδώ και μη βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν είπα. Θέτω ερωτήματα, ερωτήματα εύλογα. Διότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλεκόμεθα στη συζήτηση αυτή και θέτουμε τα ερωτήματα αυτά. Σε ένα επικοδομητικό πνεύμα τονίζω. Η κατάσταση θα πρέπει να εξεταστεί και τι κάνουν ακριβώς οι Ρώσοι, αλλά το train and equip πού υπήρξε αποτελεσματικό. Αν υπήρξε αποτελεσματικό, ας κάνουμε κι άλλο τέτοιο. Αλλά αυτό που βλέπω είναι μια τεράστια επένδυση και πάρα πολλές ανοιχτές ερωτήσεις. Η CBST λόγω της συζητήσεως και λόγω και λόγω της ε, έντονης συζήτησης της κάπου την οδηγήσαμε και υπήρξαν και στοιχεία μετριασμού του κινδύνου μέσα σε αυτήν την... Ε, και γι' αυτό υπάρχουν και άλλα, τα, άλλα project τα οποία χρηματοδοτούνται. Και βεβαίω η επανεξέτασή του είναι πολύ δύσκολη από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι είναι λοιπόν φυσιολογικό να θέτει κανεί ερωτήσει χωρί ε, να αναγκαστεί κανεί να χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμού του είδου η νευρισιά, η στρατιωτική, οι ένοπλε δυνάμει και τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τέτοια. Και τα ξαναλέω αυτά διότι εδώ δεν είναι πλέον business as usual. Ορίστε κύριε Νταμζόν. Έχω μία ερώτηση. Πού είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει train and equip, πού ακριβώς κάνει train and equip, δηλαδή εκπαίδευση και εξοπλισμό. Απάντηση. Το να δίνετε εξοπλισμό, πολεμεφόδια και όπλα, είναι αυτό train and equip. Train and equip, δηλαδή εκπαίδευση και εξοπλισμός έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση training mission, αλλά δεν έχουμε train and equip και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει equip το 2013 και μετά το 2016 δύο ε, εκπρόσωποι ξεκίνησαν την ιδέα του Train and Equip, που έτσι γράφεται κιόλα και στα έγγραφα του Συμβουλίου, διότι δεν είχαμε το τμήμα του, το οποίο ακόμα δεν έχουμε το τμήμα του εξοπλισμού. Και μου ομιλείται για τη CBST. Μπράβο η CBST. Και εγώ συμμετείχα στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο για την CBST. Καταλήξαμε να μην επιτρέπεται να δώσουμε πυρούνια στις ενόπλε δυνάμει, διότι απαγορευόταν να δοθεί οτιδήποτε το θανατηφόρο και ένα πυρούνι θεωρήθηκε ότι μπορεί να είναι θανατηφόρο. Ωραία, είναι θεμητά τα ερωτήματα, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια άλλη ατζέντα από πίσω και η ατζέντα αυτή είναι ότι δεν θα πρέπει να αγγίζει τα θέματα της ασφάλειας και τα στρατιωτικά θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά είναι τα θεμελιώδη τα οποία ταράσσουν τη συζήτηση αυτή. Και αυτό που με ενοχλεί είναι που κάνετε δίκη προθέσεων. Πρόκειται για δίκη προθέσεων. Δεν υπάρχει πρόγραμμα ε, εκπαίδευση και εξοπλισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε λοιπόν να επικρίνετε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν λειτουργεί το τρένο που είπα αφού δεν υπάρχει. Εάν υπήρχε θα μπορούσε κανεί να το αξιολογήσει. Το μόνο που κάναμε είναι να πούμε ότι δεν υπάρχει τμήμα equip για να συμπληρώσει το πρόγραμμα train. Αυτή είναι η ιδέα του CBSD και του συμπληρώματο που θέλουμε να κάνουμε. Όπου δηλαδή κάνουμε εκπαίδευση ε, στρατιωτικών δυνάμεων να μπορούμε να κάνουμε και εξοπλισμό. Γιατί ξαναλέω, στο συμπιεστή δεν υπάρχει τίποτε το θανατηφόρο. Απολύτω τίποτα. Και φτάσαμε μέχρι σημείο ε, να του στερούμε και εξοπλισμό που βεβαίω δεν είναι θανατηφόρο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή για να φωνεύσει κάποιο έτερον. Ορίστε, αυτή είναι η διαφορά. Μιλώ για train and equip, διότι η πρόταση λέει train and equip. Δεν μιλώ για το CBST. Αυτό συζητώ. Είναι θεμητό, είναι η απάντηση αυτή τώρα, είναι ε, ε, θεμητό να σκεφτεί κανείς, βλέποντας τη συμπεριφορά αυτών των στρατιωτικών απέναντι στους πληθυσμούς των χωρών τους, τι θα κάνουν εάν τους δώσετε και εξοπλισμό. Και για το G5 Sahel είδαμε ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα αναλάβει τα ενία Ευρωπαϊκή Ένωση ω διαμαγεία, θα λυθούν τα προβλήματα. Η Ένωση πρέπει να γνωρίζει πού πάει να μπλεχτεί. Γιατί μπορείτε να δείτε και άλλε χώρε τι κάνουν και πώ λειτουργήσαν τα δικά τους ε, συστήματα. Νομίζω ότι κάνουν πολλές υποθέσεις και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε. Θα βάλετε το σήμα τη Ένωσης ε, Φαδιά πλατιά πάνω στον εξοπλισμό. Μα επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Δίκη προθέσεων η απάντηση του κ. Ντανζόν. Είναι, δεν μπορούν δηλαδή να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν μπορούν να δώσουν εξοπλισμό σε ενόπλε δυνάμει μια τρίτη χώρα, διότι αυτομάτω θα τα κάνουν αυτά χωρί να λάβουν καμιά προφύλαξη ή απολύτω αρνητικά. Τι είδου κριτική είναι αυτή, και σε βάρο των χωρών μελών. Διότι λέτε ότι δεν λειτουργήσε όταν τον ανέλαβαν οι χώρε μέλη. Και φαντάζομαι ότι η δική μου χώρα, η Γαλλία, θα είναι πάνω-πάνω στον κατάλογό σα ότι κάνουν ό,τι θέλουν δηλαδή. Ακούστε, δεν ανέχομαι να διεξάγεται δίκη προθέσεων συστηματικά στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και στις χώρες μέλη. Να υπάρχουν προφυλάξεις, να υπάρχουν ρήτρε προφύλαξης, έλεγχοι. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ ποτέ δεν είδα σε 10 χρόνια που είμαι Ευρωβουλευτής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιου είδους αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς να υπάρχει τέλος πάντων κάποια πρόβλεψη για πλαισίωση, εγγύηση και ούτω Ποτέ δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο λοιπόν διεξάγεται αυτή η δίκη προθέσεων σήμερα. Να υπάρχει έλεγχος ασφαλώ. Γι' αυτό κάνουμε και ε, έκθεση και πρόκειται να τροπολογήσουμε και Άρα να ξεκινείτε με μια τέτοια ε, προκατάληψη ότι πάμε να βάλουμε τα δάχτυλα σε ένα μηχανισμό που θα τα καταστρέψει, τα δάχτυλα ή το μηχανισμό, αυτά νομίζω ότι είναι απολύτω εκτό θέματο. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταμουζόν. Εσεί θέλετε να απαντήσετε ακόμη μια φορά. Κοιτάξτε, το μόνο που, το πρώτο που μπορώ να κάνω είναι να ε, ξαναπώ τα όσα είπα στην αρχή. Ότι έχουμε πολλέ ερωτήσει, όχι όμω του ίδιου που είπατε ανέφερα τα αφηγήματα και τα συνέδεσα με ερωτήσει που συνδέονται με τη σειρά του με μια πολύ σημαντική συζήτηση για το πώ θα γίνει η αξιολόγηση του κινδύνου, πώ ε, θα διαμορφωθεί η συνοχή, ποια μέτρα κατά τη διαφθορά θα ληφθούν, ώστε να παραμείνει σε υγιή πλαίσια η συζήτηση, όπου να μην απευθύνουμε οι μεν χαρακτηρισμού του δε. Ας διεξαχθεί μια συζήτηση η οποία θα στρέφεται γύρω από τα πραγματικά ερωτήματα και νομίζω κάτι τέτοιο θα είναι υγιές. Αντί, ξαναλέω, να εκτοξεύουμε χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Ιδού. Εσείς κύριε Μπουσέρ. Ναι, για την ερώτηση του τι πρόβλημα προσπάθουμε να λύσουμε. Οι τζιχαντιστές ε, προσέξαν τον Παμάκο και υπήρξαν κάποιες ε, ε, δυνάμεις ασφαλείας και βοηθήσαμε με, την, με το μηχανισμό ειρήνης για την Αφρική και στην Σομαλία και τις ομαλικές ε, στρατιωτικές δυνάμεις ε, βοηθήσαμε που τώρα ανακτούν τον έλεγχο της χώρας και παρότι δεν είναι τέλεια η κατάσταση ανακτήσαμε σε μεγάλο βαθμό την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα αυτή οπότε υπάρχουν περιστάσεις όπου υπό την απειλή βίαιων ε, ενοπλών ομάδων είναι δύσκολο να αποκαταστήσει κανείς την ειρήνη αν δεν έχει ανθρώπους ένοπλους. Και τώρα αναγνωρίζετε ότι η προϋπόθεση για κάθε ανάπτυξη και άνθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επαρκής αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας σε μια χώρα. Κύριε Ντονζό, αναφέρατε το παράδειγμα των Ρώσων που παρενέβησαν ε, γιατί η Ευρωπαίοι δεν έκαναν πολλά ε, και στη Σομαλία ε, η υποστήριξη και η εκπαίδευση δεν μπόρεσε να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειαστήκαμε να πάρουμε ανθρώπους από τη Σομαλία, τους μεταφέρουμε στην Ουγγάντα και υπήρχε ανάγκη. Εκεί χρειάστηκε να εξοπλιστούν με, με ε, άρβιλα και με ε, ρούχα αγκαρίας και λοιπά, στολές και τα λοιπά, για να συνεχίσουν. Υποστήριξη λοιπόν των εκπαιδευόμενων κληρωτών, αυτά αναλύθηκαν τελικά από τις ΗΠΑ. Εκεί ήταν, έλαβαν οι Αμερικανοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε. Εξαρτιόταν 100% από τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική για την νέα εκπαιδευτική αυτή αποστολή. Όσον αφορά τι εγγύσει που έχουμε, κυρίω αφορούν σε οποιαδήποτε δράση ασφάλεια που χρειάζεται απόφαση από το Συμβούλιο και μάλιστα ομόφωνη των 28 Υπουργών. Και αυτό αποτελεί εγγύηση ότι τα πράγματα αυτά λαμβάνονται σοβαρός υπόψη. Όσον αφορά την ίδια την πρόταση και τις εγγύησεις κατά της κατάχρησης των όπλων, η ιδέα δεν είναι να δοθούν χρήματα στα, σε τρίτα μέρη για να προμηθευτούν εξοπλισμούς μόνους, μόνοι τους η European Peace Facility θα προβλέπει ότι θα χορηγείται ο εξοπλισμός από χώρες μέλη, ίσως όπλα και πολεμεφόδια, ίσως όχι. Κυρίως θα πρόκειται για τηλεπικοινωνιακό υλικό και μεταφοράς προσωπικού. Η ιδέα δεν είναι τόσο να δοθούν χρήματα σε μια τρίτη χώρα ώστε αυτή να προμηθευτεί τον εξοπλισμό η ίδια. Η ιδέα είναι να απευθυνθεί η Ένωση σε χώρα μέλος η οποία θα εξαγάγει ή οδήποτε στρατιωτικό υλικό μετά από απόφαση του Συμβουλίου γιατί για να γίνει αυτό χρειάζεται να δοθεί άδεια εξαγωγής από μια χώρα μέλος του εξοπλισμού και κάποια χώρα μέλος θα αναλάβει το καθήκον να εφαρμόσει την σχετική δράση που θα συνίσταται στην παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού. Η πρόταση προβλέπει ότι το τρίτο αυτό μέρος που μπορεί να είναι χώρα μέλος εννοώ θα εφαρμόσει την δράση στήριξης τρίτης χώρας στη, βάση σύναψης συμφωνίας που θα πρέπει να περιλαμβάνει και την υποχρέωση και των δύο πλευρών και του τελικού δικαιούχου. Επομένω, να διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι δίνει εγγυήσει σχετικά με τη χρήση του στρατιωτικού εξοπλισμού. Επιπροσθέτω, προβλέπονται διατάξει για ελέγχου από ανθρώπου που διορίζει η European Peace Facility και αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους μεταξύ άλλων και για την χρήση του εξοπλισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα, πληρωθεί, δεν θα, δεν ο εξοπλισμός αυτός, ούτε θα δοριστεί σε παραπέρα ε, άτομα ή φορείς. Αυτά έχουν βεβαίω, για τα πράγματα αυτά οι χώρες μέλη έχουν ιδιαίτερε ευαισθησίε. Η ιδέα πάντως είναι ότι δεν θα δώσουμε είτε χρήματα σε τρίτη χώρα για να αγοράσει όπλα η ίδια και πολεμεφόδια και να κάνει μετά ό,τι θέλει με αυτά, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ενδιάμεσο πιθανότατα χώρα μέλο για να παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό και για να ελέγχει για ποιου λόγους, για ποιου σκοπούς χρησιμοποιείται ο εξοπλισμό αυτός. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο σύντομο. Και Χάκμαν, παρακαλώ. Ε, κύριε Χάουτμανς, ναι, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ε, καθυστέρησα λίγο να έρθω, αλλά ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για κάτι νέο, ίσως λίγο τολμηρό και ο, ο, ο κόσμος έχει ερωτήσεις διότι πρόκειται για κάτι νέο. Είμαι πεπισμένη όμως ότι είναι απαραίτητο, όχι αναγκαίο μάλλον θα λέγω, όχι απλά χρήσιμο ως μέσο. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Ντανζό, πρέπει όλοι να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να εγγυηθούμε τον έλεγχο σε όλα αυτά τα μέρη. Αλλά ακούμε διάφορε επικριτικές ερωτήσει, Αυτό είναι κομμάτι τη δημοκρατία. Αλλά ξέρετε, στην πράξη θα αποδειχθεί η χρησιμότητα. μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα εφόσον χρησιμοποιηθεί καλά αυτό ο μηχανισμό. Και θα πρέπει να διαπιστώσουμε, αυτό το διαπιστώσουμε εφόσον δούμε καλά αποτελέσματα επί τόπου. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε πότε θα δούμε ορατά αποτελέσματα από αυτό το Ταμείο ε, Επιτόπου. Κάτι τελευταίο. Έγιναν πολλές ερωτήσεις και πιστεύω ότι υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα του μηχανισμού, αλλά το ερώτημα είναι γιατί το Συμβούλιο ε, φέρει τόσες επιφυλάξεις. Όπως είπατε αγαπητή κυρία, εάν ο κόσμος ε, το εμπιστεύεται και εμείς πρέπει να τους πείσουμε το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Εγώ δεν μπορώ να τους πείσω ε, αν δεν χρησιμοποιήσουμε ε, το κονδύλι αυτά επί τόπου και δεν φέρουμε καλά αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε τι επιχείρηματα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε το Συμβούλιο να φέρει θετική γνωμοδότηση για τον μηχανισμό αυτό. Ευχαριστώ. Is somebody Θέλει κάποιος να απαντήσει. Εγώ επιχειρήματα δεν μπορώ να σας δώσω προς υποστήριξη του μηχανισμού. Αλλά όπως λέτε το ότι όλα αποδεικνύονται, αποδεικνύουν τη χρησιμότητά του στην πράξη, αυτό συμβαίνει σε, πολλές, σε πολλά πράγματα. Αλλά δεδομένων των δεσμεύσεων που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και για λόγου συνοχή, δεν υπάρχει λόγος ένα εργαλείο σαν αυτό να μην περιλαμβάνει έναν καλό μηχανισμό λογοδοσία, αναθεώρηση των προγραμμάτων που θα υποστηριχθούν, εάν χρειαστεί να τα προσαρμόσει ανάλογα με τι συνθήκε. Γιατί ξέρουμε ότι στι χώρε αυτέ τα πράγματα αλλάζουν σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι ο σκοπό μα, όχι όλα τίποτα. Αλλά πρόκειται για κάτι καινούριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συστήματα αναθεώρησης και λογοδοσίας δεν θα ισχύει για αυτό εδώ γιατί μιλάμε για κάτι νέο. Αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορούμε να έχουμε τι διασφαλίσει που έχουμε και σε άλλου τομεί και να δούμε πώ μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό ή αν θα χρειαστεί να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο. Αλλά το να τα αφήσουμε έτσι τα πράγματα είναι ακόμη πιο θολά. Αν μπορέσουμε να καθορίσουμε σωστά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια θα πείσουμε περισσότερο και τον κόσμο. Ευχαριστώ. Κύριε Μπουσέ, ένα λεπτό. Θέλω και εγώ να κάνω μια ερώτηση, ε, κύριε Μπουσέ. Μιλάμε για τρίτες χώρες. Μιλάτε και για Ουκρανία και αυτήν περιλαμβάνεται στις τρίτες χώρες. Yes, please. To the last question, Κοιτάξτε, για την τελευταία σας ερώτηση δεν υπάρχει γεωγραφικός αποκλεισμός, γεωγραφικός περιορισμός. Αν διαβάσετε δηλαδή τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, βεβαίως κυρίως δίνουν έμφαση στην Αφρική, δέχτηκαν όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός. Αν λοιπόν αποφασίσει το Συμβούλιο, μπορεί να αναλυφθεί δράση και υπέρ της Ουκρανίας. Υπάρχουν βέβαια ιδιαίτερες ευαισθησίες εκεί λόγω τη ιδιαίτερη γειτονία τη με μια συγκεκριμένη χώρα αλλά θα μπορούσε η European Peace Facility να χρηματοδοτήσει και τέτοια δράση υπέρ της Ουκρανίας. Όσον αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας εισηγήτριας, συμφωνούμε ότι χρειάζεται έλεγχος του μηχανισμού Πρόκειται για CFSP, για ΚΕΠΑ δηλαδή. Επομένως αυτό τον πυλώνα της ε, πρόκειται για κοινοτικό πυλώνα. Επομένως, Χρειάζονται αποφάσει για κάθε δράση και μάλιστα ομόφωνα από το Συμβούλιο. Υπάρχει Επιτροπή των Χωρών Μελών που εγκρίνει το σχετικό προπολογισμό και βεβαίω έχουμε και εκθέσει και για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο. Εμπλέκεται δηλαδή και το ελεγκτικό συνέδριο και όπω είπα προηγουμένω, η ιδέα είναι να και προβλέπεται κιόλα να υπάρχουν ελεγκτέ οι οποίοι θα πηγαίνουν επί τόπου για να ελέγξουν όχι μόνο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των χωρών μελών, αλλά και για το τι γίνεται με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Εάν γίνεται δηλαδή η χρήση του σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής της Ένωσης και ιδίως όσον αφορά σεβασμό ανθρώπινων δικαιωμάτων, ε, ειρήνη, σταθερότητα κλπ. Για την ερώτησή σας πώς μπορείτε να το πλασάρετε αυτό στις χώρες μέλη. Οι υπουργοί έχουν γνώση του ότι ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90 ας πούμε όταν άρχιζαν τα πράγματα αυτά να κινούνται. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Μέρη στα οποία ταξίδευσα ως νέος δεν θα μπορούσα να πάω τώρα. Και οι πολίτες γνωρίζουν ότι ο κόσμος έχει γίνει πια επικίνδυνος και η European Peace Facility υποτίθεται θα δώσει την ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ποτέ να μπορεί να δρά σε καταστάσεις που έχουμε γύρω, γύρω μας με όλα τα μέσα. Ε, αν έτσι κρίνουν οι χώρες μέλη και μάλιστα ομόφωνα. Και επειδή ακριβώ είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αξίε και αρχέ και πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ., είναι καλύτερα να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό και να έχει την ικανότητα, να δοθεί η ικανότητα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θα δοθεί έτσι η βεβαιότητα στους πολίτες ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για να αντιμετωπίζει την καταστάση στο μέλλον και με σεβασμό στις αρχές της. Αυτό θα έλεγα στους πολίτες. Χωρίς βεβαίως να είμαι βουλευτής, έτσι δεν είναι. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα έχετε καλύτερα επιχείρηματα. Ευχαριστώ κύριε Μπουσέρ. Ευχαριστώ επίσης και την προσκεκλημένη μας. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, που εγώ τη βρήκα τουλάχιστον προσωπικά πολύ χρήσιμη. Και πριν να τελειώσω, έχω κάποιες παρατηρήσεις. Σχετικά με το ιστορικό αυτού του θέματος ΤΡΙΑ και πρώτα η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, που είναι η 15η πρώτου του 19, 12 το μεσημέρι. Έτσι δεν είναι, κυρία Χάουτμαν. Έγκριση στην ΑΦΕΤ 21η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Αυτό λοιπόν ήταν το ζήτημα 3. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την και τον προσκεκλημένο μας. Το επόμενο σημείο. Αποκινούμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα συζητήσουμε την κατάσταση ασφαλείας στην Αζωφική θάλασσα και στα στενά Κέρτσα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν μέχρι τις 4 η ώρα. 12 λεπτά διάλειμμα. Thank you very much. Thank you very much.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

Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, επιτρέψτε μου να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας. Το επόμενο σημείο σημερίσια διάταξη είναι η κατάσταση ασφαλείας στην Αζωφική και στα στενά του Κέρτς. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ τους ξένους μας, τους προσκεκλημένους μας. Σούμπερ κυρίως, επικεφαλής ε, του τμήματος κύριος Σέλ, επικεφαλής ε, ε υπεύθυνο για τη Ρωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ, στο επιτελείο του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ολεξίλ Μακέλεβ, πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ουκρανίας και Αμάντα Πάουλ, υπεύθυνη για το, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Πριν από ένα μήνα είχα τη δυνατότητα να, την ευκαιρία να συμμετάσχω στην επίσκεψη της, ε, στη Μαριούπολη και στην ε, Αζοφική, μαζί με την Υποπιτροπή Άμυνας. Αφέτα. Στις 25 Νοεμβρίου ε, δύο κρανικά πλοία, σε δύο κρανικά πλοία έγινε επίθεση από την Ρωσία και επιτέθηκαν σε έξι Ουκρανούς ε, στρατιώτες και 24 ε, συνελήφθησαν. Και μετά από αυτό ο κύριος Ποροσέγκο είπε ότι είναι αναγκαίο να κηρυχθεί ο στρατικό νόμος στην Ουκρανία σε διάφορες ε, περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πολύ δυσχερής και μια περαιτέρω, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή αυτή. Μπορούμε, πιστεύω, να συνεχίσουμε στη συζήτηση με τα μέλη του πάνελ και τους ε, ευρωβουλευτές μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό σας προτείνω να δώσουμε 5 7 λεπτά σε κάθε ομιλητή και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μακέγεφ από την Ουκρανία. Παρακαλώ, έχετε 5 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και θα ήθελα ξεκινώντας να επενέσω την Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα αυτό της Μαύρης Θάλασσας κοντά στα στενά του Κέρτς γιατί πράγματι η κατάσταση στην Αζωφική ε, και ευρύτερα στην ε, Μαύρη Θάλασσα αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύθραυστη και το γεγονός ότι η δική σας ε, επιτροπή ασχολείται για τρίτη φορά με το θέμα αυτό και το γεγονός ότι επισκέφθηκε μάλιστα πρόσφατα την Ουκρανία προκειμένου να πληροφορηθεί από τις ε, Ουκρανικές αρχές για την, και τις τοπικές αρχές για την κατάσταση που κρατεί εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και αυτή τη στιγμή η κατάσταση ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί διεθνώς. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που συμπεριλάβα το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή σας. Ε, επιτρέψατε μου να σας περιγράψω συντομία το τι συνέβη. Ε, τρία ουκρανικά πλοία ε, μετέβαιναν από το ένα λιμάνι στην ε, ακτή της Μαύρης Θάλασσας προς την Αζωφική, προς τη Μαριούπολη. Ήταν μια στάνταρ ρουτίνα ανάπτυξη δυνάμεων, κάτι συνηθισμένο για οποιοδήποτε ναυτικό. Ε, τα, η ομάδα αυτή ήταν ε, μικρή, δεν υπήρχαν πλέον όπλα και ενώ ε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας προσεγγίζοντας την ακτή ειδοποίησαν την εκτοφυλακή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στον ρωσικό μύθο, ο οποίος λέει ότι η Ουκρανία δεν είχε το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο ότι διέπραξαν μια παραβίαση, μια, έκαναν μια πρόκληση. Αλλά τι είδου ε, παραβίαση ήταν ε, αυτή. Ε, αυτό είναι εντελώ ασαφές. Καταρχήν, το, τα ρωσικά ε, υδάτινα σύνορα δεν ε, παραβιάστηκαν ούτε νόμιμα ούτε παράνομα. Γιατί το 2014 η Ρωσία ε, κατέλαβε και προχώρησε στην προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ε, σύνορα, δεν υπάρχει ζώνη των 12 μιλίων γύρω από την Κρυμαία όπως ισχυρίζονται οι Ρώσοι. Αυτό δεν ευσταθεί. Και βεβαίως αυτό συμφωνεί με την ε, Σύμβαση των Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Η ελεύθερη ναυσιπολογία εδώ επιτρέπεται από την διεθνή νομοθεσία. Άρα η προσωρινή κατάληψη της Κρυμαίας από τη Ρωσία δεν αλλάζει αυτή την κατάσταση. Και η, επίσης η διμερή συνθήκη του 2003 η οποία εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, ορίζει την αζωφυθική και τα στρενά του Κέρτς ως ε, εσωτερικά ύδατα και το άρθρο 3 της συνθήκης επικυρώνει ότι όλα τα πλοία της Ουκρανίας, στρατιωτικά ή εμπορικά, έχουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοεία στην ζώνη αυτή και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, και αντί να τους ε, παράσχει την, να εκπληρώσει την υπηρεσία ελέγχου, η Ρωσία ε, προσπάθησε να εμποδίσει την διέλευση των Ικρανικών πλοίων και παρέλειψαν να ενημερώσουν ε, το κέντρο, τα κέντρα ναυσπλοείας στην ε, Ισπανία κάναμε επανελμένους ελέγχους, δεν έγινε τέτοιου είδους επίσημη γνωστοποίηση ότι είχαν κλείσει τα στενά του Κέρτς. Οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις ε, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και στρατιωτικών ε, ε, αεροπλάνων αποστάλησαν εκεί και προσπάθησαν να μπλοκάρουν τη διέλευση των Ουκρανικών πλοίων προχωρώντας σε επικίνδυνους χειρισμούς. οι περαιτέρω εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα ποιος ε, προκάλεσε την πρόκληση. Βλέπουμε την απρόκλητη επίθεση στα ουκρανικά πλοία σαν μια ενσυνείδητη πράξη επίθεσης εκ μέρους της Ρωσίας. Ε, τα δικά μας πλοία αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ουκρανικό λιμένα της Οδυσσού, στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά στη συνέχεια η Ρωσία άρχισε να τα ακολουθεί και να τους επιτίθεται με όπλα τα ουκρανικά πλοία δεν άνοιξαν πυρ σε απάντηση της ρωσικής επίθεσης. Άρα λοιπόν ε, δεν αξιολογήθηκε σωστά η σοβαρότητα της κατάστασης καθότι η Ρωσία ε, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια κατέλαβε, προέβη στην κατάσχεση τριών ουκρανικών πλοίων σε αυτή την ε, ζώνη των υδάτων. Ήταν απολύτως ε, ξεκάθαρο από τις συστήσεις που έγιναν ότι η επίθεση δεν έγινε στα ουκρανικά πλοία, δεν έγινε αυθόρμητα, αλλά ήταν μια ενσυνείδητη πράξη επίθεσης κατά της ε, Ουκρανίας, ε, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Ρωσία ε, στην, περιοχή είναι να κλείσει την Αζωφική θάλασσα και για την Ουκρανία και για τη διεθνή ναυσιπλοεία με τον τρόπο αυτό ε, θανατώνοντας την οικονομία της ακτογραμμής της Αζωφικής στην Ουκρανία και δημιουργώντας στρατιωτικές προϋποθέσεις για μια επίθεση κατά της Ουκρανίας από τη θάλασσα. Σαν ε, αποτέλεσμα όλων αυτών η Ουκρανία ήταν αναγκασμένη να απαντήσει προκυρήσοντας ε, την ε, κατάσταση έκτακτης, το νόμο στην περιοχή αυτή παρακαλώ να κατανοήσετε ότι είναι ένα αμυντικό μέτρο που έχει σαν σκοπό να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε καλύτερα για περαιτέρω στρατιωτικές προκλήσεις εκ μέρους της Ρωσίας. Οι, ανθρωπιστικοί, ε, οι ανθρωπιστικές συνέπειες για την ε, ρωσική της στην περιοχή ή έχει δραματικές επιπτώσεις. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 17 Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη φυλακή της, στις φυλακές της Ρωσίας. Υπήρχαν μέχρι στιγμής, τώρα έχουμε 24 ε, εχμαλώτους πολέμου που η Ρωσία αντιμετωπίζει ως εγκληματίες πλέον και τους έστειλαν από την υποκατάληψη τελούσα Κρυμαία στη Μόσχα και όλες αυτές τις μέρες δεν είχαμε απολύτως καμία δυνατότητα να αποκτήσουμε ε, πρόσβαση στα, στους ναυτικούς μας. Ούτε καν οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, ούτε ο Ερυθρός Σταυρός, ούτε ε, εκπρόσωποι άλλων διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι το αίτημά μα. Ζητούμε από την ε, Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να παρέμβει στο θέμα αυτό και να αποκτήσει πρόσβαση στους ε, εχμαλώτους ε, πολέμους. Ε, συγγνώμη. Και θα ήθελα να τελειώσω απευθύνοντα μια σημαντική έκκληση προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνοντας τις ευχαριστίες μου θα ήθελα να εκφράσω το αίτημα μιας περαιτέρω υποστήριξης προς τη δική μας ε, πλευρά σε σχέση με την ε, ρωσική επιθετικότητα στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, εμείς χαιρετήσαμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ασοφική τον Οκτώβριο. χαιρετήσαμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και προτείνουμε τα μέτρα τα οποία προτάθηκαν να περάσουν σε πρακτική εφαρμογή. Καθώς η κατάσταση στην Αζωφική επιδεινώνεται, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν συνιστά μόνο θέμα ασφαλείας για την, Ουκρανική, ε, για την Ουκρανία, αλλά μια μίζωνη πρόκληση για την Ευρώπη και την Ευρωτολαντική ε, Συμμαχία. Και πάλι θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να καταγγείλετε αυτή την ε, πράξη ρωσικής επιθετικότητας και να καλέσετε τη Ρωσία να την ε, τερματίσει. Επίσης θα πρέπει να ζητήσετε από τη Ρωσία να απελευθερώσει τους κρατούμενους. τα στρενά του Κέρτς θα πρέπει να είναι ανοιχτά στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, στα ουκρανικά πλοία και στα ευρωπαϊκά πλοία, στα πλοία με ευρωπαϊκή σημαία, τα οποία θα πρέπει να έχουν μια ελεύθερη πρόσβαση στην αζωφική. Επίση, θα ήθελα να σε απευθύνω μια έκκληση να εξασφαλίσετε η Ρωσία να ε, αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις ε, πράξεις της. Και ένα σημαντικό εργαλείο εδώ είναι η επιβολή κυρώσεων εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Ρωσία προς τα λιμάνια της και εκείνους που είναι υπεύθυνοι για αυτό το συμβάν. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις αυτές ε, και σας ευχαριστώ και για αυτές τις εκκλήσεις που απευθύνατε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ντίρκ Σουμπέλ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρότι θα προτιμούσα να ήταν πιο ευχάριστη η περίσταση. Ο κύριος μακιέφα ανέφερε την ουσία της όλης υπόθεσης, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Να αναφερθώ στη δική μας αντίδραση, στο ότι πιστεύουμε ότι συμβαίνει εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ε, ε, και εκ μέρους της είπα εκπροσώπου, σύμφωνα με τη δήλωσή της της 28 Νοεμβρίου, εκφράσαμε μια παγιά θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Συνολικά υπήρξαν τρεις ε, παγκόσμιες δηλώσεις με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την δήλωση του εκπροσώπου μετά από το περιστατικό στις 26 Νοεμβρίου με τα όπως ανέφερα και εγώ υπήρχε η δήλωση των 28 με πλήρη συμφωνία και των 28 και μετά συμμετείχαμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δήλωση των G7 επίσης σημαντική δήλωση των σημαντικότερων χωρών του κόσμου. Την παρουσία στιγμή θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να δείξουμε όλοι ε, προσοχή ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση τη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα έχουμε όλοι εκφράσει τι βαθιέ μα ανησυχίε για την κατάσταση. Ήταν κάπω αναμενόμενο ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν προ αυτή την κατεύθυνση και φυσικά όλα αυτά είχαν ως αφετηρία την ε, οικοδόμηση της γέφυρας ε, στο Κέρτς. Είχαμε όλοι εκφράσει την ανησυχία μας ε, για την κλιμάκωση των εντάσεων στα στενά του Κέρτς και στην Αζωφική θάλασσα που όπως μας είπε ο κύριος Μακέιεφ οδηγήθηκε στην κατάσχεση των ε, πλοίων, ε, τους πυροβολισμούς, ε, τη σύλληψη των στρατιωτικών. Όλο αυτό λόγω της απαράδεκτης στρατιωτικοποίησης της περιοχής εμείς απευθύνουμε έκκληση για αποκλιμάκωση αναμένουμε ότι η Ρωσία θα ελευθερώσει χωρίς όρους ε, τα πλοία και τα πληρώματά τους. Οι συλληφθέντες, ναύτες, ναυτικοί και οι τραυματισμένοι θα πρέπει να λάβουν αμέσως ε, την αρρωγή και την υποστήριξη που χρειάζονται. Δεν γνωρίζουμε μάλιστα ποια είναι η κατάσταση των τραυματιστέντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τη Ρωσία ότι θα διασφαλίσει περαιτέρω την ε, ανεμπόδιστη διέλευση από την Αζωφική θάλασσα σύμφωνα με το Διεθνέ δίκαιο και με, το διμερές, ε, με τη διμερή συμφωνία που έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά και που χορηγεί ελεύθερη πρόσβαση στα ρωσικά και στα ουκρανικά πλοία. Αυτή τη στιγμή, όπω γνωρίζουμε, σύμφωνα με τι δικέ μα πληροφορίε, τα πλοία που κατευθύνονται προ και από τα ε, ουκρανικά λιμάνια στην Αζωφική θάλασσα δεν επιτρέπεται να διέρχονται από τα στενά του Κέρτσα, από τη ρωσική εκτοφυλακή. Αυτό περιλαμβάνει και κάποια ε, πλοία με ε, σημαίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία σε πολλές ε, στη λιμάνια ουκρανικά της περιοχής και σε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες. Όπως είπε, είπε ότι εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πρόσφατα, πριν κλιμακωθεί η κατάσταση, τα περιστατικά στην Αζωφική θάλασσα αποδεικνύουν πως η αστάθεια και οι τάσεις εντείνονται όταν υπάρχει παραβίαση των βασικών κανόνων της διεθνούς συνεργασίας μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Η οικοδόμηση της γέφυρας Κέρτ, όπως είπα προηγουμένω, ε, πραγματοποιήθηκε χωρίς συνένεση της Ουκρανίας και αποτελεί άλλη μια παραβίαση της Ουκρανικής ε, ε, εδαφική κυριαρχίας και ακεραιότητας. Χρειάζεται αποστρατικοποίηση της Αζωφική θάλασσας και να επιτραπεί η ναυτική κυκλοφορία στα στενά και στη θάλασσα. Διότι τώρα δυστυχώ μπορούν από τη γέφυρα να περάσουν μόνο πλοία ενό συγκεκριμένου μεγέθου, γιατί νομίζω έχει ύψου μόνο 33-34 μέτρα ε, η γέφυρα και μόνο μικρότερα πλοία από αυτό μπορούν να περάσουν από τα στενά. Ενώ αυτό δεν συνέβαινε προηγουμένω. Τώρα, όσον αφορά τη, στρατιωτικοποίηση τη Αζωφική θάλασσα, πιστεύουμε ότι δεν συμφέρει κανέναν. Δεν κάνει τίποτα παρά να αποσταθεροποιεί την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα. Να επαναλάβω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρω την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα τη Ουκρανία με τα διεθνώς αναγνωρισμένα τη σύνορα. Δεν αναγνωρίζει την παράνομη προσάρτηση της Κρημαϊκής Χερσονήσου από τη Ρωσία. Δεν χρειάζεται να πω, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελπίζουμε ότι τα αιτήματά μας που έχουμε εκδώσει εμείς με τις δηλώσεις μας θα ικανοποιηθούν από τη Ρωσική Ομοσπονδία η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κλείσω, και στο επίπεδο της ύπαρξη της εκπροσώπου και Προέδρου κυρίας Φεντερίκα Μογκερίνη υπήρξαμε σε επαφή με διάφορους εταίρους από τότε που ξεκίνησε η κλιμάκωση και θα συνεχίσουμε τις επαφές με σκοπό να συνεργαστούμε ε, στενά με τους διεθνείς μας εταίρους σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σούμπερ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ρομπέρτ Ψέλ. Παρακαλώ. Να ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό εδώ καθόμαστε ένα δίπλα στον άλλο. Κύριε Σούμπελ, ε, εσεί εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ τον ΝΑΤΟ. Αλλά αυτά που θα σα πω τώρα δεν θα διαφέρουν από αυτά που ακούσαμε, γιατί οι θέσει των οργανισμών μα ε, επί του ζητήματο αυτού είναι παρεμφερεί, όπω και πρέπει να είναι. Για όσους δεν ε, παρακολουθήσατε λεπτομερώς, να σας πω ποια ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στη χρήση ε, στρατιωτικής δύναμης από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας ε, στην Αζωφική θάλασσα. Πρώτα απ' όλα χρονολογικά είχαμε μια δήλωση από τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ. Την επόμενη μέρα ο Γενικός Γραμματέας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ποροσέγκο και συμφωνήθηκε ότι το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία θα συστήσουν μια έκτακτη συνάντηση της ε, Επιτροπής ε, ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που έλαβε χώρα την ίδια μέρα. Και το ΝΑΤΟ ως βορειοατλαντικό σύμφωνο με τη συμμετοχή και των 29 ε, συμμάχων εκδόθηκε μια δήλωση. Θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης είχαμε μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού τον κύριο Παραβέ και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας στην συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στο ζήτημα. Είχαμε μία σειρά υπουργικών διασκέψεων, έχουμε μάλλον που θα αρχίσουν αύριο στο ΝΑΤΟ, είναι η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και η πρώτη συνάντηση θα γίνει με τον Γεωργιανό και τον Ουκρανό Υπουργό. Ταυτόχρονα οι συναδελφοί μου έχουν σήμερα επαφές με τους Ουκρανούς εταίρους για το ετήσιο εθνικό σχέδιο της Ουκρανίας που είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της πρακτικής συνεργασίας που έχουμε με την Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά τη δήλωση, επανέρχομαι σε αυτό. Είναι πολύ σαφής, θεωρώ. Δεδομένη της ε, χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας, οι σύμμαχοι απευθύνουν έκκληση προ τη Ρωσία να ελευθερώσει την πρόσβαση στα Ουκρανικά λιμάνια και να μην παρεμποδίζει την αυσιπλοεία που αποτελεί γεγονός, ε, δικαίωμα τη Ουκρανία. Δεν αιτιολογείται η χρήση στρατιωτική δύναμη κατά αυτών των πλοίων και, του, και των πληρωμάτων του. Και η έκκληση αυτή συνεχίζει να υπάρχει για απελευθέρωση των Ουκρανικών πλοίων και πληρωμάτων χωρί άλλη καθυστέρηση. Επίση, έγινε έκκληση για ηρεμία και προσοχή, το ΝΑΤΟ επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας και εδευκής ακεραιότητας της Ουκρανίας δεδομένων των διεθνών της συνόρων και των χωρικών της υδάτων. Καταδικάζουμε την παράνομη προσάρτηση της Κρεμαίας από τη Ρωσία, την οποία δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε και δεν αναγνωρίζουμε. Η κατασκευή της γέφυρα του Κέρτσα αποτελεί από τη Ρωσία άλλη μία παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ δηλαδή βρίσκεται με το πλευρό της Ουκρανίας και είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε πολιτική και πρακτική υποστήριξη στην Ουκρανία εντό του πλαισίου τη καθιερωμένη συνεργασία μα. Και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση. Αυτό που ανέφερε η πολιτική και πρακτική υποστήριξη. Νομίζω τα ακούσατε αυτά τα στοιχεία της πολιτικής μας θέσης. Να σας πω δύο λόγια για την πρακτική υποστήριξη. Uh, annual national program, uh, which is... Να σας αναφέρω ένα εθνικό πρόγραμμα, ένα ουκρανικό πρόγραμμα που έχουμε συζητήσει μαζί και τα πρακτικά στοιχεία της ε, υποστήριξής μας ε, ε, περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο αρρωγής, όπως είπαμε συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο ως ΝΑΤΟ όσο και ως, ως οργανισμός δηλαδή αλλά και από τους συμμάχους. Υπάρχει μια σειρά trust funds ε, για διάφορα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ε, ε, logistics, οργάνωση, ασφάλεια, στρατιωτική μετάβαση, trust fund. Έχουμε επίσης και μια σημαντική πλατφόρμα που Αναμένω ότι θα χρησιμοποιείται και περισσότερο ε, για τον ε, υβριδικό πόλεμο που διευκολύνει τη συνεργασία και εντοπίζει τις υβριδικές απειλές ε, ώστε να αναπτύξουμε αντοχή προς αυτές τις υβριδικές απειλές. Και μετά υπάρχουν και άλλα πολλά στοιχεία αυτής της συνεργασίας τα οποία είμαι βέβαιος αναμφίβολα θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω Όσον αφορά τη δική μας επιχειρησιακή παρουσία στην περιοχή, το ΝΑΤΟ μετά από την παρανοή προσάρτηση το 2014 της Κρυμαίας αύξησε σημαντικά την παρουσία του στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ε, περιπολίες ρουτίνας και ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Φέτος έχουμε πλοία του ΝΑΤΟ τα οποία πέρασαν πολύ περισσότερο χρόνο στην περιοχή 120 ε, μέρες σε σύγκριση με 80 το 2017 εδώ μιλάω για περιπολίες του ΝΑΤΟ. Φυσικά υπάρχουν και περιπολίες και παρουσία άλλων χωρών. Πολλοί σύμμαχοι αστυνομεύουν την περιοχή για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και ε, πραγματοποιούν και αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε μία βάση στην Πρέοβα. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρία μέλη του ΝΑΤΟ, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία είναι ε, ε γειτονικέ χώρε που έχουν και αυτοί τι στρατιωτικέ δυνάμει ανεπτυγμένε στην περιοχή. Υπάρχει λοιπόν ισχυρή δύναμη του ΝΑΤΟ. Εξακολουθούμε να εκτιμάμε, την κατάσταση καθώ αυτή εξελίσσεται. Θα κλείσω εδώ, αλλά ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι για το ΝΑΤΟ το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφορά πολύ ε, έναν ε, εταίρο του ΝΑΤΟ παλιό και αξιόπιστο με τον οποίο έχουμε μακροχρόνια συνεργασία. Θα κλείσω εδώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Πολ. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Θα είμαι σύντομη στις παρατηρήσεις μου, δεν έχουμε πολλά, πολύ χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό το συμβάν ήταν απολύτως ε, προβλέψιμο. Ε, το νερό έβραζε στην κατσαρόλα και θα ξεχύλιζει και είχα μια πληροφόρηση από το Think Tank μου που ανέφερε ακριβώς τις εντάσεις στην περιοχή αυτή και το, την επικείμενη κλιμάκωση. Και, αυτό το, και επίσης οι συνάδελφοι από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, τόνισαν ότι υπάρχει κίνδυνος ε, και είπαν ότι θα έπρεπε να, αποσταλεί, να υπάρξει μια διεθνής αποστολή η οποία θα μεταβεί στην ε, περιοχή εκεί για να επαγρυπνήψει. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ότι εκ μέρους της Ουκρανίας υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου, αλλά δεν θα πρέπει να υπερτιμηθεί, γιατί οι Ρώσοι προσπαθούν να το κάνουν αδύνατον για την Ουκρανία να ασκήσει τον έλεγχο στα ύδατά της. Και βεβαίως εδώ και πολλά, πολύ καιρό το Κρεμλίνο προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την ε, Ουκρανία και να εμπεδώσει την ε, κατοχή της ε, Κρυμαίας. Προδευτικά προχωρεί σε μια στρατικοποίηση της ε, περιοχής της Αζωφικής και του στόλου στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να αυξήσει την κυριαρχία των Ρώσων στην περιοχή αυτή. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν δύο στρατιωτικές βάσεις στην ε, Γεωργία και στην Αρμενία και στην ε, Συρία. Άρα πρόκειται για ένα κομμάτι ενός ε, ευρύτερου, μιας ευρύτερης προσπάθειας εγχειρήματος εκ μέρους της Ρωσίας προκειμένου να κλιμακώσει την επιθετικότητά της. Ε, όπως σας είπα, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία σοβαρή απάντηση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας που να υπερβεί τα όρια απλών δηλώσεων και εκφράσεων ανησυχίας. Ε, ε, και ε, βεβαίω υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και την Ουκρανία διότι δημιουργούνται τεράστιες επιπτώσεις στο ΑΕΠ της Ουκρανίας από τη μη πρόσβαση στους εμπορικούς λιμένες και θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτή η πρόσβαση στα στενά. Ε, Βεβαίω ο στόχος της Ρωσίας είναι κατ' ουσία να κλείσει τα στενά του Κέρτς προκειμένου να στραγγαλίσει την ουκρανική οικονομία και να ενισχύσει τη θέση της ε, Ρωσίας δημιουργώντας ένα νέο μέτωπο στην περιοχή επιπρόσθετο προς αυτό του Ντόνμπας και της, της Κρυμαίας. Πρόκειται λοιπόν για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και για να είμαι σύντομη θα ήθελα να σας δώσω μερικά παραδείγματα για πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή τη συγκυρία εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας. Καταρχήν, ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές να μιλάμε για επιβολή κυρώσεων, αλλά πέρα από την διατήρηση των κυρώσεων που ήδη επευλήθηκαν το Σεπτέμβριο στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, πιστεύω ότι εάν αυτή η προσπάθεια στοχίσει θα πρέπει να υπάρχει υπάρξει ένα πέρασμα σε στοχεσμένη επιβολή κυρώσεων για τις ε, παραβιάσεις αυτές και για την, ε, ευρύτερα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δοκιμάτων στην ε, Κρυμαία. Σαν δεύτερο σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση του Άντριου Βίλσον σε σχέση με την ανάπτυξη μιας διεθνούς ναυτικής αποστολής στην Αζωφική και στα στενά του Κέρτς, οι Ουκρανοί ε, κατηγορούν τη Ρωσία και οι Ρώσοι την Ουκρανία. Άρα μια διεθνής αποστολή εκεί θα μπορούσε να προλάβει μια περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Όσον αφορά το ρόλο του ΝΑΤΟ, συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ενισχύσει ε, την παρουσία του εκεί. Έχει, το έχει ήδη κάνει, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και ίσως να υπάρξει μια εναλλαγή των πλοίων του ΝΑΤΟ εκεί και να υπάρξουν και αμερικανικά πλοία στην περιοχή. Και ως τελευταίο σημείο, ίσως το πιο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την άμυνα της Ουκρανίας. Για αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν έχει την ικανότητα να το κάνει και θα πρέπει να τους δώσουμε ε, πυραυλικά συστήματα στην, ε, για τα πλοία. Eh, Ωραία κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, δηλαδή στα τσέχικα. Θα αξιοποιήσω τη δυνατότητα που μου δίνετε ως ε, πρόεδρος. Πριν δώσω τα λόγια, το λόγο σε άλλα μέλη της Επιτροπής μας, των Επιτροπών μας δηλαδή, για να με ακριβείς, θα θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι προς τον κύριο Σούμπελ. Κύριε Σούμπελ, μου φαίνεται ενδιαφέρον που κανένας από εσάς δεν έχει χρησιμοποιήσει τη σωστή λέξη που έπρεπε να χρησιμοποιούμε σε τέτοιες ε, καταστάσεις. Δηλαδή να μιλήσει, δεν μίλησε κανείς ε, για υπεριαλισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη σωστή ορολογία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι θα γίνει όσον αφορά τις κυρώσεις. Εγώ πηγαίνω συχνά στο Ντομπάς, ε, συζητώ με εκπροσώπους του στρατού, με θελοντές, ε, με μάχημους ε, και διάφοροι μου λένε «Εσείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πλάκα μας κάνετε». Θα χαθεί εμπιστοσύνη προς την Ουκρανία για να ε, ε, που, που έχουν εκρανεί σε εμά. Θα πρέπει να μαχηθούμε για να διατηρήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξή, κύριε Σιουμπέλ. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πιο αυστηρές οι κυρώσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις προς όλα τα μέλη της Άνω Βουλής του Ρωσικής Ομοσπονδίας που ενέκρινε την είσοδο των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι θα είναι μια εντυπωσιακή κίνηση τέτοιου είδους κύρωση. Και μετά ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν θα μπορούσαμε ως κύρωση για μια τέτοια κατάσταση να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ρωσικών πλοίων στα λιμανιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτέ οι ερωτήσεις είναι για τον κύριο Σούμπαλ. Και μετά έχω άλλη μία ερώτηση, αν προλαβαίνουμε, προς τον κύριο Ψτσέλ. Και τώρα θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Η κυρία Μούδη νομίζω θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. And, uh, Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ απόψε το απόγευμα και πραγματικά αυτό δείχνει την σοβαρότητα με την οποία ασχολείται η Επιτροπή με το θέμα αυτό. Ε, πιστεύω ότι κάτω από το πρίσμα των όσων πόθηκαν για την διασύνδεση μεταξύ Γεωργίας και Ουκρανίας, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ε, το πρώτο ερώτημα είναι ε, σχετίζεται με τα όσα συνέβησαν το 2008 στην Γεωργία και ίσως ε, ε, οι ανεπάρκειες ε, τότε διευκόλυναν, διευκόλυναν τόσα συνέβησαν στη συνέχεια στην Ουκρανία. Θα ήθελα να μας πείτε με περισσότερες λεπτομέρειες τι φοβάστε σε σχέση με την στρατηγική δράση. Το δεύτερο θέμα αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές. Ε, μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν οι κυρώσεις. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και βεβαίως, ε, όπως ακούστε, υπάρχουν ε, και, υπάρχει και το αίτημα για περισσότερες κυρώσεις. Σε σύστημα, με είπε και, και η κυρία Πάουλ. Επιπλέον, αναφέρθηκε μια αποστολή ε, παρατήρησης της ε, ναυσιπλοείας στην ε, περιοχή εκεί, των θαλασσών. υπάρχουν κάποια σχετικά πλάνα, υπάρχει κάποια προετοιμασία προκειμένου να ξεκινήσει μια τέτοια αποστολή. Τέλος, τα όσα υπόθηκαν σε σχέση με τα συμβάντα στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, θα μπορούσατε να μας πείτε αν υπήρξε και μία αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλατε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω για την αντίδραση της Γερμανίας στην έκκληση του κυρίου Ποροσέγκο όσον αφορά την υποστήριξη για την Αζωφική θάλασσα. Και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω οι Ουκρανικές αρχές ε, πώς αποτιμούν την κατάσταση όσον αφορά την αντίδραση των συμμετεχόντων της Συμφωνίας του Μίνσκ ε, όσον αφορά την όλη κατάσταση. Ποια είναι η δική τους αντίδραση. και τι άλλες εκκλήσεις έχουν ε, υπάρξει, τι άλλα αιτήματα έχουν ε, ακούσει από τις Ουκρανικές αρχές για τη Γερμανία και τα άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Harms. Ευχαριστώ κύριε Χάρμς, έχετε το λόγο. Thank you. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που γίνεται η παρούσα συνάντηση γιατί απογοητεύτηκα μετά από τη διάσκεψη κορυφής G20 στη Βραζιλία χωρίς κανένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Πούτιν μετά από την δημόσια δήλωσή του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει μόνο όταν ο Ποροσένικο δεν θα είναι πλέον πρόεδρος της Ουκρανίας. Εγώ τουλάχιστον αυτό το πράγμα το βρήκα συγκλονιστικό ως δήλωση. Το ίδιο όπως και την πρόσφατη σύγκρουση στα στενά του Κέρτς. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ στο θέμα αυτό δεν θα πρέπει να φανούμε πολύ αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Οι ερωτήσεις μου απηχούν και αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Εξ όσων γνωρίζω, η εντολή του ΟΑΣΕ της ε, αποστολής παρακολούθησης καλύπτει και την θάλασσα του Αζόφ, την Αζοφική θάλασσα και τα στενά του Κέρτς. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και ρωτώ, γιατί κανείς δεν προετοιμάζει μια τέτοια επέκταση εφόσον αυτή χρειάζεται. Δεύτερο, παρουσία του ΝΑΤΟ. Διαβάσαμε τα νούμερα σχετικά με αυξημένη στατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Μαύρη Θάλασσα. Δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό να υπάρξει ξεκάθαρη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή αυτή του κόσμου όπου σημειώνονται τα προβλήματα, δηλαδή στη θάλασσα του Αζόφ και στα στενά Κέρτσε. Τελευταία ερώτηση, λίγο διαφορετική, αφορά περισσότερο τις εξελίξεις στην ίδια την Ουκρανία και ειδικότερα στην Μαριούπολη, η οποία αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο προβλήματα λόγω του αποκλεισμού. Και ούτως ή άλλως είναι μια πόλη που αντιμετωπίζει πολιτικά προβλήματα. Μια ασταθή κατάσταση που εμφανίζεται ξανά και ξανά και η κατάσταση αυτή γίνεται όλο και πλέον ασταθής εφόσον οι οικονομικές προοπτικές γίνονται όλο και πιο αδύναμες. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι παραπάνω για να σταθεροποιήσει την Μαριούπολη, να είναι ας πούμε πλέον παρούσα στην Μαριούπολη. Υπάρχουν σχέδια της Ουκρανικής κυβερνήσεως επ' αυτού. Τελευταία ερώτηση. Η αναβολή των τοπικών εκλογών. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα και πότε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρμς. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων Πρώτο γύρο λοιπόν απαντήσεων αν ε, δεν έχετε αντίρρηση. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Πρώτα, Μούντι, η απάντηση της Γεωργίας και η αδύναμη περί την Κρυμαία. Είναι αυτά που δίνουν αφορμή στο ρωσικό καθεστώς. Δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας. Εάν δηλαδή θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στεναρά στις προκλήσεις. Διδαχθήκαμε από αιώνες γειτονίας προς την Ρωσία και τα χρόνια βέβαια της Ουκρανικής ανεξαρτησίας ότι η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της δύναμης και πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται μαζί της μόνο με αποδύναμη, από αποθέσεως ισχύω. Μάθαμε επίσης σήμερα ότι ο όρος κυρώσεις δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, δυστυχώς, εδώ στις Βρυξέλλες και σε πολλές άλλωστε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σας παρακαλώ όμως να αντιληφθείτε ότι είναι και το μόνο ειρηνικό μέσον που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι για να ανακόψουν τις ε, ρωσικές στρατιωτικές δράσεις και επιθετικότητα. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Ουκρανοί στρατιωτικοί, στο μέτωπο, που είναι παραπάνω από 400 χιλιόμετρα μέτωπο απέναντι στους Ρώσους. Και βλέπουμε τώρα και μια επιθετική δράση και στην θάλασσα. Άρχισαν το 2014 οι Ρώσοι και τώρα επεκτείνουν την επιθετική τους δραστηριότητα και στη θάλασσα. Ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γι' αυτό οι κυρώσεις είναι πολύ σημαντικές. Και αυτό θα έλεγα και στον κύριο Γιούρεκ και στην κυρία Χάρμς. Εξετάστε το θέμα των κυρώσεων. Απαγόρευση πρόσβασης στα ρωσικά λιμάνια, Ρόκανο και Διέιτς. Απαγόρευση σε ρωσικά σκάφη που έρχονται από αυτά τα λιμάνια να μπουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια και προσωπικές κυρώσεις κατά εκείνων οι οποίοι διέταξαν τις δράσεις αυτές από τον ρωσικό πολεμικό στόλο. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο των κυρώσεων. Κύριε Γιούρεκ, ρωτήσατε για την δράση της Γερμανίας και αν αυτή συζητήθηκε. Πράγματι, ο πρόεδρος μου αμέσως τηλεφώνησε στην Ομοσπονδιακή Καγκελάριο τη Δευτέρα νομίζω και την παρακάλεσε να παρέμβει. Ο ίδιος προσωπικά το έχω συζητήσει στο επίπεδο των πολιτικών διευθυντών το λεγόμενο Normandy Format την προηγούμενη Δευτέρα και είχαμε και επίσημη απάντηση από τους φίλους μας ε, της Γερμανίας και Γαλλίας οι οποίοι καταδίκασαν την επιθετικότητα της Ρωσίας. Αυτές τις καταδίκες οφείλουμε τώρα να τις μεταφράσουμε σε ενέργεια, σε δράση. Εκεί βλέπω εγώ ανάγκη ηγετικής ε, στάσης των Ευρωβουλευτών. Τώρα, η αποστολή του ΟΑΣΕ, πράγματι η ειδική αποστολή παρακολούθησης, του ζητούμε να παρακολουθούν και να συντάξουν ειδική έκθεση. Γνωρίζετε ότι στον ΟΑΣΕ οι δυνατότητες μας είναι κάπως περιορισμένες, διότι είναι οργάνωση η οποία βασίζεται στη συνένεση. Η δε Ρωσία δεν θα επιτρέψει επέκταση της εντολής της. Αλλά αυτό είναι που θα έπρεπε ωστόσο να κάνει η διεθνής κοινότητα. Να πιέσει δηλαδή τη Ρωσία να το δεχτεί. Τώρα οι εξελίξεις στην ίδια την Ουκρανία και οι υποδομές στην Αζωφική θάλασσα, κυρία Χάρμς. Αυτό αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να σκεφτεί σχετικά τα πράγματα αυτά και να μας ε, υποστηρίξει στην δημιουργία τις αναγκαίες υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου ο άμαχος πληθυσμός υφίσταται τα δεινά και οι ρωσικές δυνάμεις αποκλείουν λιμάνια, το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ζημία στο εθνικό προϊόν της Ουκρανίας και ειδικότερα της περιφέρειας αυτής. Άρα, επενδύσεις σε έργα υποδομής γύρω από την Μαριούπολη και βέβαια ενίσχυση των αμυντικών μας ικανοτήτων. Αυτό βεβαίως απευθύνεται ως έκκληση προς το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τους, και τις συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό σε διμερή βάση. Αναβολή των τοπικών εκλογών, κυρία Χάμς. Αυτό προβλέπει ο στρατιωτικός νόμος. το προβλέπει η στρατιωτική νομοθεσία και η Κεντρική Επιτροπή Εκλογών μας ενημέρωσε περί της αναβολής των εκλογών. 30 ημέρες προβλέπει ο στρατιωτικός νόμος. Ευχαριστώ που μου δώσατε και πάλι το λόγο λοιπόν και ελπίζω ότι επίνησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ο κύριος Σίμπελ, ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Ας ξεκινήσουμε από την ερώτηση της κυρίας Χάρμς από το τέλος. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για τη Μαριούπολη ως πόλη και τις, γύρω, και τις λοιπές περιοχές εκεί τριγύρω. Ήδη κάνουμε πολλά. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15 εκατομμυρίων, ολοκένουργιο για την αναζωογόνηση της Ουκρανίας, όπως το ονομάζουμε. Και ενώ εμεί συζητάμε εδώ, αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο συζητείται στη σχετική ομάδα το ίδιο πρόγραμμα μεταξύ άλλων. Αυτό φυσικά πριν από την κλιμάκωση στην Αζωφική θάλασσα. Απλά να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει την αποκέντρωση, τη διακυβέρνηση, την οικονομική ανάκαμψη και ειδικά για τη Μαριούπολη αφορά την αποκέντρωση τη δημιουργία ενό περιφερειακού κέντρου εκπαίδευση προσωπικού στη Μαριόπολη. Επίση, μάλιστα, έχουμε χρηματοδοτήσει το φωτισμό των δρόμων στην πόλη. όπω ξέρει όλος ο κόσμο η πόλη αυτή είναι στην, Ανατολή της Ουκρανίας, στην Ανατολική Ουκρανία και εξυγχρονίστηκε και είναι πολύ όμορφη τώρα. Επίσης, ε, αποκαταστήσαμε κρίσιμα δίκτυα παροχή ε, νερού και ε, υποδομέ υδροδότησης σε όλη την περιοχή. Θα σα δώσω και περισσότερε πληροφορίε, αν θέλετε διμερώ. Επίσης αυτό το πρόγραμμα των 15 εκατομμυρίων έχει ε, πέραν αυτού υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για την τοπική οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο του προγράμματος αποκέντρωσης και βελτίωσης της πόλης και της διοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Καταπολέμησης Διαφθοράς. Όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά με διάφορους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας. Αυτά είναι κάποια πράγματα που κάνουμε ήδη και που προτιθέμεθα να κάνουμε και φυσικά ευχαρίστως να εξετάσουμε και άλλα ενδεχόμενα. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσο η Ουκρανία θα συμπεριληφθεί στον OCSMM, εγώ είχα συναντηθεί με το ΕΣΥ και μου είπαν ότι καλύπτουν τη Μαριούπολη αλλά όχι τη θάλασσα. Οπότε χρειάζεται επιπλέον εντολή. Και όπως είπε ο κύριος Μακέη, Χρειαζόμαστε συμφωνία όλων. Αλλά όπως είπε ο κύριος ε, Μακέ, δεν θα είναι εύκολο να λάβουμε το πράσινο φως από όλους και ειδικότερα από ένα κράτος μέλος του ΟΑΣΕ. Για το ζήτημα τώρα των κυρώσεων ε, και εγώ πήγα μετέβη δύο-τρεις φορές στην περιοχή στην Ανατολική Ουκρανία, στο Σύροκ, ε, στην περιοχή των Συράξεων και είναι θλιβερό το όσο βλέπει κανείς εκεί. Ε, οπότε έχω την ίδια αίσθηση και με εσάς ότι έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα. Αλλά δεν μπορώ εγώ να λάβω εδώ δημοσίω κάποια απόφαση. Το Συμβούλιο πρέπει να λάβει τη σχετική απόφαση ε, με ομοφωνία και των 28 κρατών μελών για τυχόν περαιτέρω κυρώσει. Απλά ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά την δήλωση που έκανε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος στην τελευταία της πρόταση και το είπα ήδη και στην παρέμβασή μου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι αποφασισμένη να δράσει ανάλογα σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους. Τι σημαίνει αυτό σε περίπτωση που δεν απελευθερωθούν τα πλοία, τα πληρώματα, η ναυτική σύντομα από τις ρωσικές αρχές. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα τι αποφάσεις θα ληφθούν, αλλά σας διαβεβαιώ ότι το παρακολουθούμε στενά και θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ε, δηλώσω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο. Κύριε, κυρία Πόλ. Θα είμαι πολύ σύντομη για τη Γεωργία. Ναι, θεωρώ ότι ήταν ε, τεράστιο σφάλμα η μη απόκριση την εποχή εκείνη γιατί στείλαμε ένα μήνυμα προς, τους, ε, προς τη Ρωσία ότι θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν και το τίμημα είναι πολύ χαμηλό. Και αυτό τους εθάρρυνε να κάνουν ό,τι έκανα στη συνέχεια. Ε, δεν μπόρεσαν λοιπόν να αποτραπούν ε, οι Ρώσοι, να αποτραπεί η ρωσική επιθετικότητα. Και θα πρέπει να επιβληθούν και οι Ρώσεις για αυτή τη στιγμή ε, για τη Ρωσία βεβαίως η στρατηγική του στόχη είναι πολύ πιο σημαντική από τις ε, δίποτε ε, κυρώσεις. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, η αστάθεια στη Μαύρη Θάλασσα είναι φιάλτης για την Τουρκία και η Άγκυρα είναι σε επαφή τόσο με τον Ποροσέγκο όσο και με τον Πούτιν. Και ο Ερντογάν προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο. Βεβαίως, στο παρελθόν η Τουρκία δερμάτισε ένα χρήσιμο ρόλο ε, ε, διευκολύνοντας την απελευθέρωση των Τατάρων κρατούμενων από την Κρυμαία αλλά τι θα γίνει τώρα εκ μέρους της Τουρκίας, αυτό που μένει να το δούμε. Βεβαίως υπάρχει το δυναμικό μιας απόκρισης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος για το τι πρέπει να γίνει, γιατί αυτή είναι μια ε, γλώσσα ο ε, όρος συμπεριαλισμός είναι κάτι το οποίο ανάγεται στο παρελθόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο διεθνές ε, δίκαιο και πιστεύω ότι τα όσα έγιναν δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει. Το ΝΑΤΟ είναι δύναμο, λέγεται, αλλά παρόλα αυτά μετά το πέρος του μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου, ε, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Αύριο ο κύριος Μακεύ μαζί με τον Υπουργό Κιμκίν θα συναντήσει 29 υπουργούς των συμμάχων χωρών του ΝΑΤΟ και θα συζητήσουν σχετικά. Βεβαίως ε, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω ότι το ΝΑΤΟ έχει την ε, εντολή αυτή τη στιγμή τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τις διάφορες χώρες να συνδράμουν την Ουκρανία. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω συνδρομή και ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, καλύπτονται από την κοινή δήλωση την οποία ε, εξάδωσε το ΝΑΤΟ και την στηρίζουν ξεκάθαρα. Έχω μια επιπρόσθετη ερώτηση. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία με πυρομαχικά και όπλα. Απάντηση. Αν αυτός είναι ο τύπος, η μορφή βοήθεια ε, που χρειάζεται η Ουκρανία, αυτό είναι απόκειται στις ε, αρμοδιότητα των χωρών ε, μελών να το αποφασίσουν. Η Ουκρανία δεν βρίσκεται, δεν προλαμβάνεται σε καμία μαύρη λίστα όσον αφορά την διεθνή νομοθεσία. Άρα εναπόκειται στην ευχαίρεια της κάθε χώρας συμμάχου εταίρου της Ουκρανίας να το πράξει και έχει πολλούς εταίρους η Ουκρανία εντός του ΝΑΤΟ. Ε, είναι, και... είναι 5 και 5. Σας ευχαριστώ όλους. Θα πρέπει τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα η κυρία Μούντι να αναλάβει τώρα την Προεδρία.

Yeah. Ο πρόεδρος κύριος Μακάλιστερ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω το, ε, τη μεγάλη χαρά να μπορώ να σας υποδεχτώ στην παρούσα συζήτηση για την επιρροή της Ρωσίας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Έχουμε και την Κλέρ Μούντι ως, ε, που αντικαθιστά την κυρία Φωτίγκα ως αντιπρόεδρος της ΣΕΝΤΕ. Γνωρίζετε ότι οι νοτιοανατολικοί γείτονέ μα, ε, ιδίω οι έξι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων που πορεύονται προ την ένταξη στην Ευρώπη μέσα από μια μακρά και δύσκολη πορεία, φέροντα ε, την κληρονομιά του παρελθόντο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ προσφέρουν με την ένταξη στου οργανισμού αυτού μια προοπτική ασφάλεια και σταθερότητα. Υπάρχουν ωστόσο κακεντρεχεί έξωθεν επιρροέ με στόχο να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Θα, θα ρίξουμε ιδιαίτερο φως σήμερα στην επιρροή της Ρωσίας. Βέβαια είμαι βέβαιος ότι οι προγνώμονές μας θα εξετάσουν το ε, ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή επίσης και επιρροή Τουρκίας, χωρών του Περσικού κόλπου, Κίνα και του βασικού μας εταίρου των ΗΠΑ. Με συμβουλές και παροχή βοήθειας υπό όρους, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει το όραμα της μελλοντικής ένταξης, αλλά ταυτόχρονα ζητεί μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με τους κανόνες, ενώ το Κρεμλίνο όχι. Προσπαθεί να ενθαρρύνει αντιδυτικά αισθήματα, να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών αυτών, χρησιμοποιώντας ε, και ανοιχτά και ε, κρυφά μέσα και όσο γνωρίζουμε, οι soft power operations του Κρεμλίνου χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, οικονομική επιρροή, ε, κρίσιμες ε, υποδομές, πολιτική επιρροή μέσω ισχυρών ε, ηγετών, χρηματοδοτήσεις κομμάτων και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά και με την υποστήριξη των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η μεγαλύτερη ζημιά που κάνει η Ρωσία είναι με το να σπέρνει τη διχόνοια και βασισμένη σε εθνικούς εξτρεμισμούς μεγεθύνοντας υφιστάμενες διαφορές, ξεκινώντας νέες διαφορές, προωθώντας συγκρούσεις και ανακόπτοντας μεταρρυθμίσεις και την δημοκρατική πορεία. Για παράδειγμα, η προσπάθεια να υπονομεύσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, ένα παράδειγμα παραπληροφόρησης και χρήσης στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στην Ελλάδα που προσπαθούν εκεί να προωθήσουν εθνικές διαφορές κατηγορώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρόνο σε αυτήν για να ασχοληθεί με τα θέματα της, ε, των Δυτικών Βαλκανίων και με την προοπτική που έδωσε, αλλά έχουν καθυστερήσει τα πράγματα αυτά και έχουν οδηγήσει σε μεγάλη απογοήτευση για τις ε, δυτικές χώρες των, ε, μάλλον για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η ε, σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει, γιατί να χάνει τη μάχη για να κερδίσει τις καρδιές και τα πνεύματα των ανθρώπων εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα της Ρωσίας. Χρειάζεται αντίδραση στη ρωσική επιθετικότητα θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε το καθήκον μας, θα πρέπει να κρατήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια υψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων μας, να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για μεταρρυθμίσεις προενταξιακά και ταυτόχρονα συμφιλίωση, ισχυρή δικαιοσύνη, ισχυρή οικονομία, ανεξαρτησία και ανταγωνιστικότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μαζί με τις προσπάθειες των πρωτεύουσών μας πρέπει να μην φυστούν προσπαθειών για να επιτρέψουν να αποκτήσουν ανθεκτικότητα οι δημοκρατικοί θεσμοί των χωρών αυτών, να κλείσουν τα κενά της παραπληροφόρησης και να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση. Αυτά από την πλευρά μου. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Κλέρ Μούντι για να κάνει εισαγωγικέ παρατηρήσει και αναμένω μετά να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με του προσκεκριμένου μα. Σα ευχαριστώ, David. Πράγματι, πολλά από τα όσα θα έλεγα τα είπατε ήδη. Θα αρκεστώ λοιπόν να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που συμπροεδρεύω στην παρούσα ε, συνεδρίαση. Έχω παρόμοιες ανησυχίες ε, γύρω από τα Δυτικά Βαλκάνια που κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην ρωσική εξωτερική πολιτική, χωρίς απαραίτητα να είναι προτεραιότητα στις εξωτερικές τους υποθέσεις. Όπως ελέγχει όμως, υπάρχει ιστορικά δημοτικότητα, έντονη δημοτικότητα των Ρώσων στην περιοχή αυτού του κόσμου και έχουν και μια χαμηλού κόστου στρατηγική για να αυξήσουν την επιρροή τους εκεί. Και βέβαια να εκμεταλλευτούν κάποιες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αργή πρόοδο της εξέλιξης των σχέσεων εκεί. Θα προχωρήσω λοιπόν στο να σας παρουσιάσω τους συνομιλητές μας. Πρώτα θα ήθελα να απευθύνω το καλό ορίσατε στον κύριο Μπέρτσεφ, ο οποίος θα συζητήσει την ε, Foreign Policy Agenda των Ρώσων και τις επιπτώσεις και εκεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Research Fellow στο Κέντρο Σλαβικών και Ανατολικοευρωπαϊκών ε, Μελετών στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και Senior Fellow στο Ατλαντικό Συμβούλιο. Ορίστε, αν θέλετε, κύριε Μπέτσεφ. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση. Η Ρωσία βρίσκεται στα μυαλά όλων. Ακούσαμε για τη συμφωνία των Πρεσπών και είναι εντυπωσιακό σε αυτή τη συμφωνία ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα κράτος μόνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που παραδοσιακά συνεργάζεται με τη Ρωσία, τώρα αντιτίθεσε αυτήν. Μας δείχνει πως η Ρωσία έχει κάνει φίλο στην περιοχή αλλά και τους έχει χάσει και που βρίσκεται η ρωσική επιρροή σήμερα. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα. Θα είμαι σύντομος. Θα σας δώσω μια γεύση των όσων προσπαθεί η Ρωσία να κάνει και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Δύση για το πώς ε, προωθεί ουσιαστικά. Να σας προωθήσω και εγώ λίγο τον εαυτό μου, σας διαφημίσω λίγο τον εαυτό μου, το βιβλίο μου ε, που αφορά ακριβώς τη Ρωσία. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι η Ρωσία έχει επιστρέψει στην περιοχή. Μετά από την Κρυμαία φυσικά η Ρωσία είναι πολύ πιο ορατή. Αλλά αυτό είναι λίγο λάθος ε, θα έλεγα. Η Ρωσία δεν έχει φύγει ποτέ από τα Βαλκάνια, δεν είχε φύγει από τα, Βαλκόνια, από τα Βαλκάνια. Ε, ε, δραστηριοποιείται στην περιοχή με διάφορου τρόπου μέσα στα χρόνια μετά από την κατάρρευση τη ε, Σοβιετική Ένωση. Τη δεκαετία του 90 είχαμε τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και η Ρωσία προσπάθησε να γίνει ένα από του διαμεσολαβητέ με αμφίβολη επιτυχία αλλά μετά ο Πούτιν αποφάσισε ότι δεν είχε νόημα αυτό το εγχείρημα και σταμάτησε την δραστηριοποίηση στη Βοσνία και στο πέδιο της Ρωσίας. Αυτό ήταν το πρώτο. Μετά τη δεκαετία του 2000 η Ρωσία ε, ανακάλυψε ότι μπορούσε να είναι η υπερδύναμη ενεργειακή στην περιοχή και ότι τα Βαλκάνια ήταν μια περιοχή διέλευσης. Και μετά είχαμε την κρίση της Ουκρανίας. Εκεί θα έλεγε κανείς ότι η Ρωσία ήταν και ανταγωνίστρια αλλά και εταίρος για τη Δύση. Για έργα όπως το South Stream, όσο και αν ήταν επίμαχα, αυτά είχαν να κάνουν και με τα Δυτικά Βαλκάνια και τις ανάλογες εταιρείε και οι αντιδράσει ήταν μεικτές. Ε, η Ρωσία ε, δεν δημιούργησε πολλά προβλήματα τότε όπως σήμερα. Και σήμερα τι γίνεται σε αυτή την τρίτη φάση. Οι Ρώσοι δεν έχουν θετική ατζέντα, δεν θεωρούν ε, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι χώρο επιρροής τους, ούτε τη Σερβία, ούτε οποιονδήποτε άλλο. Δεν του βλέπουν ως πιθανούς ε, συμμετέχοντες στην Ευρασιατική Ένωση. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να ζημιώσουν τη Δύση όσο το δυνατόν περισσότερο. Θεωρούν τα Δυτικά Βαλκάνια είναι η αχίλιο πτέρνα της Δυτικής Συμμαχίας όπου μπορούν να υποκινήσουν ε, ταραχές ε, και να αποκομίσουν κάποιο γεωπολιτικό πλέον έκτημα και φυσικά έχουν ένα αφήγημα το οποίο αιτιολογεί τις δράσεις τους κατηγορούν τη Δύση ότι έχει αναμειχθεί στην αυλή τους, σε χώρες της επιρροής τους, ε, της πρώην επιρροής τους, Μολδαβία, Γεωργία κτλ. Και ενοχλούνται που όλο και περισσότερες από αυτές τις χώρες στρέφονται πλέον προς τη Δύση. Οι Ρώσοι Ε, δίνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ το δικό του φάρμακο ουσιαστικά. Τώρα, προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα των γεγονότων, αλλά τις σκέψεις των Ρώσων. Ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν κάποιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα, κάποιο διαπραγματευτικό χαρτί. Συχνά τη Ρωσία τη βλέπουμε ως ανταγωνιστή και αυτό δίνει στον Πούτιν την εντύπωση ότι έχει κάποιο κύρος. Η Ρωσία δεν είναι τόσο σημαντική για τις οικονομίες της περιοχής, αν εξαιρέσουμε την ενέργεια. Δεν έχει στρατεύματα επί τόπου, όπως το ΝΑΤΟ. ούτε συμμετέχει στις κοινωνίες ε, των δημοκρατών της προηγουσλαβίας, όπως ε, η Δύση. Αλλά στην πραγματικότητα έχει κάποια επιρροή και ε, θέλει να αποκομίσει και κάποια κέρδη από όλη αυτή την εμπλοκή της. Γιατί έχει τόσο επιτυχία η Ρωσία στην περιοχή συχνά. Σκεφτόμαστε ε, ότι οι δραστηριότητες του Κρεμλίνου υποκινούνται από τη ρωσική κυβέρνηση, από την, elite, ε, από την οικονομική ελίτ της Ρωσίας και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την πολιτική, αλλά και τη ζήτηση επιτόπου στην περιοχή. Υπάρχει αυτή η άλλη πλευρά δηλαδή. Κοιτώντα τα Βαλκάνια, εκεί υπάρχουν πολύ πιθανοί εταίροι για τους Ρώσους, ξεκινώντας από τις πολιτικές ελίτ, που πολύ συχνά παίζουν το πλέον καθιερημένο παιχνίδι της εξισορρόπησης ε, δυνάμεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας ουσιαστικά το ανέφερε κάποιος πολιτικός ως ε, το να κάτσε σε δύο καρέκλες. Ε, άνθρωποι δηλαδή που προσπαθούν να αποκομίσουν γεωπολιτικά ωφέλη μέσω μια συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά και ερχόμενοι εδώ στι Βρυξέλλε για να λάβουν ε, παραχωρήσει από τη Δύση. Διότι διαφορετικά θα πέσουν πάλι στα δίχτυα τη Ρωσία. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίω επιχειρηματίε στι κρατικέ εταιρείε ενέργεια, για παράδειγμα, που για διάφορου λόγου του συμφέρει το status quo διότι δημιουργεί κάποια κέρδη τα οποία μπορούν να μοιραστούν και με τη Ρωσία και σε μέρη όπως η Σερβία σε κάποιο βαθμό η Μακεδονία και το Μαυροβούνιο και σίγουρα η Ρεπούμπλικα Σέρψκα υπάρχει μια ευνοϊκή ε, κοινή γνώμη προς τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποια εθνικιστικά κινήματα κόσμος που ξανασυζητά τα δεκαετία του 90, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, ε, το κοσυφοπαίδιο. Θεωρείται η Ρωσία ως αντίβαρο προς τη Δύση, ειδικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό οι Κωσοβάριο, ότι οι Μαυροβόνοι οι Μακεδόνες γνωρίζουν τη Ρωσία καλά, δεν μιλούν την ρωσική γλώσσα, δεν κατανοούν πολύ καλά τη ρωσική κοινωνία, την ιστορία και ούτω καθεξής αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι αφού η Ρωσία είναι εχθρός των ΗΠΑ ε, θέλουν να εκδικηθούν ε, τις ΗΠΑ για τον εξευτελισμό τους στη δεκαετία του 90. Και αυτό συμφέρει πάρα πολύ τους Ρώσους, ακόμη και χωρίς ε, τηλεοπτικό σταθμό, χωρίς κάποιο σημαντικό κανάλι επιρροής που να επηρεάζει το αφήγημα στην περιοχή. όπως αλλού όπου υπάρχει ρωσική τηλεόραση. Ακόμη και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, όπου παραδοσιακά η Ρωσία θεωρείται εχθρός, όπως η Αλβανία, η Ρουμανία, για να μπούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία μπήκε από την πίσω πόρτα. Φύτεψε ιστορίες ε, που δεν είναι ότι δείχνουν τη Ρωσία υποθετικό φως περισσότερο δείχνουν ε, τη Δύση ως έναν εχθρό που υπονομεύει τις παραδοσιακές αξίες των κοινωνιών που υποχρώνει τις κοινωνίες ε, να δεχθούν ε, διάφορα διάφορες διαταγές τι προσέγγισε τώρα θα έπρεπε να δείξουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ω Δύση γενικότερα στην περιοχή. Πολύ συχνά η αντίδραση σε αυτές τις εκστρατείες επιρροές είναι το να σκεφτούμε πώς θα υπερασπίσουμε τη Δύση. Αλλά εκεί υπάρχει κίνδυνος να απαντάμε στην προπαγάνδα με αντιπροπαγάνδα. Και αυτή η προσέγγιση δεν είναι πολύ επικοδομητική, ειδικότερα σε ε, κοινωνίες όπως ε, της πρώην Ιουγκοσλαβίας, όπου γνωρίζουν καλά την Δύση. Μιλάμε για μια, την Ανατολική Ευρώπη, χώρες που εντάχθηκαν ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Περισσότερο το Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τη ρωσική επιρροή, ας σκεφτούμε ε, ποιε είναι οι συνθήκε που επιτρέπουν αυτές τις κινήσεις και ποιε δράσεις Και Κλέβω τώρα λίγο από αυτά που θα πει ο Μάρκο, φυσικά ο οποίος θα τα αναλύσει καλύτερα, αλλά σκεφτείτε σε τι περιβάλλον, σε τι συνθήκες λειτουργούν οι Ρώσοι. το Κρεμλίνο χρειάζεται εκπροσώπους. Αν ο ενεργειακό τομέα ήταν πιο διαφανής, λιγότερο υποκείμενο στα κράτη, η Ρωσία δεν θα βρισκόταν σε υποσυνθήκες που τη, ευνοϊκές που τις επιτρέπουν να σφυριλατεί εταιρικέ σχέσεις συμφέροντος με τις οικονομικές ελίτ των περιοχών. Εάν τα μέσα ήταν πραγματικά ανοιχτά και όσον αφορά, υπήρχε διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μεσών μαζική ενημέρωση στην περιοχή, θα ήταν πολύ δύσκολο να φυτεύσει κανείς ψευδεί ειδήσει και να εκμεταλλευτεί τους φόβους των ανθρώπων για να προωθεί τη Ρωσία. Ή να φουσκωθεί αυτή η εικόνα της Ρωσίας ως εταίρο της δύση. Υπάρχει και αυτή η κοινωνική πραγματικότητα που πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η Ρωσία είναι εξίσου ανεπτυγμένη ε, ή μάλλον συγγνώμη, συμβάλλει το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της Σερβίας. Ενώ ο ρόλος της δεν είναι τόσο σημαντικός και τα οικονομικά ωφέλη από τη συνεργασία με τους Ρώσους είναι αμεληταία. Τα μέσα λοιπόν είναι άλλος ένας τομέας και σίγουρα το κράτος δικαίου σε μεγάλο βαθμό είναι ένα τομέα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σε όλου αυτού του τομεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο. Και εκεί μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ε, πιο εύκολο βέβαια στα λόγια παρά στι πράξει, αλλά σίγουρα αυτό είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το ΝΑΤΟ μπορεί να παίξει ρόλο στι ε, χώρε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, γιατί ε, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη Ρωσία, αλλά τελικά στη Ρωσία η εσωτερική ατζέντα, η μεταρρυθμιστική ατζέντα είναι αυτή που επηρεάζει και τη ρωσική επιρροή. Χαίρομαι που κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση εδώ και αναμένω τις ερωτήσεις και να ακούσω και τα σχόλια των υπόλοιπων ομιλητών. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάτσεφ. Uh, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάτσεβιτς, ο οποίος είναι καθηγητής ε, της ε, εφαρμογής ε, διεθνών, πρακτικής διεθνών σχέσεων ε, στο Frederick School ε, Παγκόσμιων Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και είναι πρώην πρέσβευτής του Μαυρομουνίου στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω απόψε το η παρέμβασή μου θα κινηθεί στην ίδια γραμμή με αυτή του Δημήτρη γιατί τι θα μπορούσαμε, πού θα μπορούσαμε να διαφέρουμε όσον αφορά την ε, παρέμβαση της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Ίσως θα είμαι πιο συγκεκριμένος εν σχέση με το τι κάνει η Ρωσία και πώς χρησιμοποιεί την ήπια δύναμη για να εισχωρήσει στις ε, κοινωνίες των χωρών αυτών. Καταρχήν, τι καθιστά δυνατή την άσκηση επιρροής εκ μέρους της Ρωσίας. Σίγουρα υπάρχει μια πολιτιστική εγκύτητα μεταξύ αυτών των εθνών ε, στα Βαλκάνια και της Ρωσίας και μια συγκινησιακά φορτισμένη μυθική πρόσληψη της Ρωσίας ως ε, προστάτητος δύναμης της ε, Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης η οποία αντιτίθεται στον ευρωπαϊκό δυτικό φιλελευθερισμό. Ε, δεύτερον, γιατί οι χώρες αυτές είναι ιδεώδης στόχος για τη Ρωσία, γιατί δεν έχουν πλήρως ενταχθεί ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, δηλαδή ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η Ρωσία προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και συμφωνώ τα Βαλκάνια δεν είναι μια προτεραιότητα άμεση της Ρωσίας γιατί δεν βρίσκεται στην άμεση γειτονία της Ρωσίας αλλά εάν μπορεί να αποκομίσει κάποιο κέρδος στα Βαλκάνια θα συνεχίσει να το κάνει ε, με ε, την ε, ήπια, με ένα συνδυασμό ήπιας και σκληρής δύναμης στις χώρες αυτές. Ένα τέτοιο μείγμα πολιτικής. Ποιος είναι, ποιο είναι το είδος της δύναμης που εκμεταλλεύεται η Ρωσία στα Βαλκάνια. Καταρχήν, όπως αναφέρθηκε, ήταν ε, δημοκρατικά, τα δημοκρατικά ελλείμματα των χωρών αυτών, δεύτερον οι εθνοτικές τάσεις και οι διμερείς διανέξεις ε, στα Βαλκάνια, έπειτα οι οικονομικές στρατιωτικές ανάγκες των χωρών αυτών σε ορισμένε περιπτώσεις και επίσης το αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, χρονοβόρα διαδικασία διεύρυνση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, υπάρχει ένας ε, καθρέφτης στις χώρες της Βαλκανικής όσον αφορά την κόποση για τις μεταρρυθμίσεις εκ μέρους των Βαλκανικών χωρών. Και αυτό συνιστά μια καλή ευκαιρία να παρέμβει η Ρωσία. Και έχει δύο στόχους εδώ, κατά την άποψή μου. Καταρχήν, ε, να μειώσει την επιρροή των αντιπάλων της ε, στις, ε, στην περιοχή αυτή και να παρεμποδίσει την διεύρυνση του ΝΑΤΟ και να επιβραδύνει στο μέγιστο δυνατό τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ρωσία δεν αντιτίθεται ανοιχτά στη διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να επιβραδύνει, όπως σας είπα, αυτή τη διαδικασία και να τη μετατρέψει σε μια χρονοβόρα ισοδιανικές κρεμούσα διαδικασία. Όπως είπε ο Δημήτρη, ε, οι άνθρωποι, οι χώρες, ο πληθυσμός των χωρών της Βαλκανικής δεν μιλάει ρωσικά τα τελευταία χρόνια λοιπόν η Ρωσία προσπαθεί να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα στα έψιλον ε. και υπάρχει μεγάλη ενεργητικότητα στους ε, σταθμούς ραδιοφωνίας ε, στην Σερβία, στα σερβικά. πληροφορίες που προέρχονται από τη Ρωσία. Το Sputnik είναι ο πιο δημοφιλής ρώσικος σταθμός στη Σερβία. Είναι μια εξατία λοιπόν άσκηση της ήπιας εξουσίας εκ μέρους της ε, Ρωσίας. Άρα λοιπόν εκμεταλλεύεται αυτή τα, αυτά τα δημοκρατικά ελλείμματα στις χώρες της Βαλκανικής Ρωσία και διαβρώνει ήδη αδύναμους ε, θεσμούς. Γιατί ε, υπάρχει μεγάλος ε, βαθμός διαφθοράς και προσπαθεί να διεισδύσει η Ρωσία μέσω επιχειρηματικών σχεδίων. Επίσης, Ε, προσπαθεί να επηρεάσει περιοχές όπου υπάρχουν ορθόδοξοι πληθυσμοί, όπως το Μαυροβούνιο για παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το ΝΑΤΟ ε, υπήρχε, η Ορθοδοξία, ε, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν αντίθετη στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και ήταν πολύ πιο ισχυρή από τα πολιτικά κόμματα τα οποία ήταν αντίθετα στην προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται λοιπόν τον, ορθοδεξικό, τον ορθόδοξο συγγνώμη, για να αντιταχθεί στις ε, δυτικές φιλελεύθερες ε, αξίες. Υπάρχουν λοιπόν ε, ρωσόφιλοι οργανισμοί, Ρούσκι και Μύρ και λοιπά, ο η λύκη της ε, νύχτας, ε, μια εκπαιδευμένη παραστατική οργάνωση κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι είναι δυσπαρμένοι σε ολόκληρη την περιοχή χρησιμοποιούν σαν κάλυμα για άλλου είδους ε, επιχειρήσεις διείσδυσης των υπηρεσιών της Ρωσίας στην περιοχή αυτή. Το 2016 στο Μαυροβούνιο αυτό που συνέβη είναι παράδειγμα το πώς η Ρωσία βαθμιδών διεισδύει στην κοινωνία ξεκινώντας από αυτή την ήπια άσκηση εξουσίας και προχωρώντας σε πιο σκληρά μέσα ε, που σε περιλαμβάνουν ε, υποστήριξη ε, Ρώσων των Ρώσων αξιωματούχων ε, και των ε, ρωσικών μυστικών ε, υπηρεσιών στις χώρες αυτές και τη μεγάλη αντίθεση τους στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ κύριε Γκάρτσεβιτς. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο κύριος Τσεπέρκοβιτς που θα αναπτύξει τις, τους, α, τις απόψεις του συγγνώμη, για τον ρόλο της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αναλυτής του Ινστιτούτου Στατικών Μελετών στο Παρίσι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ δύσκολο πάντοτε και ε, συνήθως ε, ομιλώ τελευταίος σε όλα τα πάνελ όπου συμμετέχω. Είναι λοιπόν δύσκολο να προβάλλω στην ομιλία μου νέες έννοιες που να μην είναι απλώς επανάληψη των όσων είπαν με τόσο φωτισμένο τρόπο οι προηγούμενοι. Θα μιλήσω τώρα για τις προοπτικές του μέλλοντος και πώς μπορεί να είναι το μέλλον όταν σκεπτόμαστε τη ρωσική επιρροή. Τα τελευταία χρόνια ρίξαν ιδιαίτερη, δώσαμε μάλλον στο Ινστιτούτο μας ε, ιδιαίτερη σημασία στην μελλοντολογία και κυρίως για να αποφύγουμε στρατηγικές εκπλήξεις στην περίπτωση της Ρωσίας δηλαδή να δούμε ποια μπορεί να είναι τα ενδεχόμενα εμπόδια και πώς να αντιμετωπίσουμε και να κατευθύνουμε τα πράγματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Για τον σκοπό αυτό δημοσιεύσαμε και πρόσφατα, δημοσίευση για το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων το 2025. Πώς δηλαδή θα είναι τα Βαλκάνια με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις νέες προκλήσεις κλπ. Η δημοσίευσή μας αυτή δεν είναι καθοριστική για το μέλλον, προβλέπει διαφορετικά σενάρια, τα οποία όμως ακόμη είναι φανταστικά. Δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μιας ευρύτατης διαβούλευσης που μας πήρε πάνω από χρόνο. Φέραμε δηλαδή μαζί ε, από εκπροσώπους κυβερνήσεων μέσω, μέχρι εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε διάφορα σημεία και στα Δυτικά Βαλκάνια και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, ώστε να έχουμε ένα είδος ευρύτατης ε, ενατένιση του μέλλοντος από διαφορετικές απόψεις. Η... Δεν θα ασχοληθώ με τη μεθοδολογία της διαβούλευσης, αλλά για να εξηγήσω πώς, τα πώς καταλήξαμε στα σενάρια. Είπαμε για τα trends, τις μεγάλες τάσεις δηλαδή, που είναι δύσκολο να αλλάξουν μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Εμείς ως ανθρώπινα όντα δηλαδή δεν έχουμε καμία σχεδόν δυνατότητα να τα επηρεάσουμε, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά Game changers, αυτά που θα αλλάξουν δηλαδή το παιχνίδι, είναι σημαντικά έτοιμοι για τη μετώπιση προκλήσεων. Αυτά τα game changers λοιπόν είναι γεγονότα ή συνθήκες οι οποίες ασκούν σημαντική επιρροή στις μελλοντικέ εξελίξεις, δηλαδή το τι κάνουμε σήμερα και από τώρα μέχρι το 2025 θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πώς ενδεχομένως θα διαμορφωθεί το μέλλον. Το καλό νέο είναι, και θα ήθελα να αρχίσω με το καλό νέο, είναι ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται το αποφασιστικότερο game changer και πρώτο στην σειρά. Και αυτό συμβαδίζει και με τα όσα είπε ο Ντίμηταρ. Η Ρωσία υπάρχει, αλλά η επιρροή τη και το πώ βλέπουν οι Βαλκάνοι το μέλλον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει τώρα να σκεφτούμε λοιπόν πώ μπορούμε ενδεχομένω να μειώσουμε τι παρενοχλήσει από τη Ρωσία. Όπω είπα, η διεύρυνση της Ένωσης είναι το game changer και είναι και ο κινητήριος μοχλός για όλες τις αλλαγές από τις δημοκρατικές μέχρι οικονομικές και βέβαια η αιρεσιμότητα παίζει και ρόλο. Ε, στη, όταν μιλώ για αιρεσιμότητα, ενώ και θετική και αρνητική αιρεσιμότητα. Άρα δηλαδή άσκηση πίεσης αλλά και οικονομική στήριξη. Κίνητρα και αντικίνητρα για να μπει μια τάξη στα Βαλκάνια. Πάντως η, η ενταξιακή διαδικασία, η οποία διαρκεί πάνω από 20 χρόνια βεβαίως, ε, επιφέρει κάποιες προκλήσεις και μια από τις προκλήσεις αυτές είναι και η αντίληψη και αυτό διαπιστώθηκε σε πολλά εργαστήρια που έγιναν σε όλα τα Βαλκάνια, είναι ότι οι άνθρωποι στα Βαλκάνια βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση καμιά φορά ως μια οντότητα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει τη σταθερότητα και την ειρήνη, αλλά με τίμημα κάποια άλλα πράγματα. Είναι δύσκολο βέβαια να το πω ε, εγώ αυτό προερχόμενος από τον οργανισμό που προερχόμαι, αλλά αυτό άλλη μια αντίληψη που πρέπει να, να αντιμετωπίσουμε, να δείξουμε δηλαδή ότι δεν βρισκόμαστε εκεί μόνο για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά και όλα τα άλλα που έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Βαλκάνια. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των βαλκανικών κοινωνιών που στήριζαν πάντοτε την ε, φιλοευρωπαϊκή πορεία και είναι το φιλελεύθερο τμήμα των βαλκανικών κοινωνιών που βλέπουν τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάποιον ο οποίος τους προδίδει εν τέλει. Και, αυτό οδηγεί σε και μάλλον αυτό πρέπει να αλλάξει σημαντικά στο μέλλον. Όπως είπα, το καλό νέο είναι ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγάλο game changer και νούμερο ένα σε όλες τις ε, συνομιλίες. Το δεύτερο νέο δεν είναι τόσο καλό. Το δεύτερο μέρος των προκλήσεων ή των game changer είναι η έξωθεν επιρροή άλλων φορέων. Και όταν μιλούμε για άλλου φορεί, οι περισσότεροι από αυτού που εντοπίζει η μελέτη μα είναι η Ρωσία πρώτη-πρώτη, η Τουρκία, οι χώρε του Περσικού κόλπου, η Κίνα και για κάποιο λόγο οι Ηνωμένε Πολιτείε μένουν απ' έξω. Στα έξι εργαστήριά μα με πάνω από 200 συμμετέχοντε, οι Αμερικανοί αναφέρθηκαν μόνο μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Κάτι ε, το οποίο μας ε, προβλημάτισε ιδιαίτερα ε, μέσα σε αυτή την έρευνα που κάναμε. Σε ό,τι αφορά την Ρωσία, έχει βέβαια την ισχυρότερη πυγμή μεταξύ όλων των άλλων εξωτερικών παραγόντων. Τη μηχανισμοί που χρησιμοποιεί για να υποσκάψει τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να παρενοχλήσει ή να αποσταθεροποιήσει θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί, οι μηχανισμοί είναι πάντα οι ίδιοι. Η Ρωσία σε μεγάλο βαθμό δεν έχει συνεκτική στρατηγική. Με την έννοια δεν προσφέρει καμιά εναλλακτική επιλογή και αυτό λέχθηκε ήδη στο πάνελ. Δεν υπάρχει δηλαδή η έννοια ότι, μάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα συγκεκριμένο στόχο, η Ρωσία όχι. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Από την άλλη μεριά, η Ρωσία συμβάλλει στην αστάθεια. Η ρωσική επιρροή προέρχεται από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι πραγματικές απόπειρες πραξικοπημάτων σε χώρες της Βαλκανικής. Θα αναφέρω μόνο ότι το 2013 έγιναν 22 κυβερνοεπιθέσεις στο Μαυροβούνιο. Το 2017 400 κυβερνοεπιθέσεις καταγεγραμμένες και συγκεκριμένη ε, επίθεση phishing με PH στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να αποφύγουν το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Δεν μιλούμε τώρα βέβαια μόνο για το Μαυροβόλιο, μιλούμε για το ΝΑΤΟ κιόλα. Η Ρωσία είναι ισχυρή στην παραπληροφόρηση. Πώ όμω, είναι απαραίτητο να κατανοήσει κανεί πώ. Ε, είναι ισχυρή ε, στο να χρηματοδοτεί news outlets, πολιτικά κόμματα, θρησκευτικέ οργανώσει. Αναφέρθηκε ήδη ο σταθμό Πούτνικ. Είναι ενδιαφέρον να δει κανεί το σλόγγαν όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014 ο Sputnik. Εμείς λέμε δυνατά αυτά που οι άλλοι θέλουν να κρύψουν. Είναι, λοιπόν, είναι ένα, σύνθημα το οποίο έχει συναισθηματική φόρτιση και είναι ξεκάθαρο. Και κυρίως σε κοινωνίες, απευθύνεται λέει σε κοινωνίες, οι οποίες αγαπούν πολύ τις θεωρίες συνωμοσία και ε, ψάχνουν να βρουν ποια είναι τα fake news κτλ. Όχι όμως τόσο. Αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τώρα, σε συνδυασμό με αυτό, δεν έρχονται δηλαδή απλώς οι Ρώσοι, δίνουν χρήματα και φτιάχνουν μια μηχανή παραπληροφόρησης. Πολλές από τις χώρες αυτές προχώρησαν και σε μεταρρυθμίσεις στα μίντια, που άλλαξαν σημαντικά την οργάνωση των, ε, ε των, του, του τύπου και προχώρησαν σε ιδιωτικοποίησεις ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες οδήγησαν να κατέχουν ραδιοσταθμούς και άλλα μίντια και σε οργανώσεις οι οποίες δεν είναι κερδοσκοπικές και όπως ο Σπούτινικ δηλαδή που εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Το βασικό αφήγημα είναι υπέρ της Ρωσίας, κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούν να επιβάλλουν τις αξίες τους. Αυτά συζητήθηκαν ήδη. Πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει και η έννοια που προσπαθούν να περάσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποσταθεροποιημένη, ε, ε, ότι βρίσκεται σε πολιτικό χάος και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέλει κανείς να ενταχθεί σε αυτήν. Στις διάφορες ε, εκδηλώσεις που διεξαγάγαμε, μας ρώτησαν γιατί να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού θα έχει πάψει να υπάρχει μέχρι το 2025. Μήνυμα το οποίο προβάλλεται συστηματικά μέσα από το ρωσικό μηχανισμό των media outlets στην περιοχή αυτή. Και τούτου λεφθέντος βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να απευθύνεται στο ε, λογικό ενώ η ρωσική προπαγάνδα στο θυμικό των ανθρώπων εκεί. Αυτή η προπαγάνδα ε, είναι ευθυνή και αποτελεσματική προσπαθεί να αλλάξει τις αντιλήψεις του κόσμου και έτσι καταλήξαμε εμείς βέβαια στα τρία σενάρια. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν, βέβαια είναι φανταστικά τα σενάρια αυτά. Έχουμε ένα πρώτο ένα φανταστικό ε, σενάριο το οποίο λέει πώς θα είναι η περιοχή αυτή το 2025. Στο πρώτο fictional σενάριο που είναι και το καλύτερο, η ώρα της Ευρώπης, προβλέπουμε μια οργάνωση από ε, ερευνητικούς δημοσιογράφους και τη λέμε Balkan Leaks, η οποία καταφέρει να δημοσιεύσει την διπλωματική αλληλογραφία από την Πάνια Λούκα στη Μόσχα με τον Ντόντε, ο οποίο είναι ε, μέλος της Προεδρίας και που ζητεί από την Μόσχα πολιτικό άσυλο εάν κάτι πάει στραβά. Θέλει δηλαδή να είναι βέβαιος ότι θα είναι ασφαλής στη Ρωσία εάν κάτι δυσάρεστο συμβεί στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό οδηγεί σε μια σειρά επεισοδίων και καταλήγει αυτός να αναγκαστεί να καταλήψει την εξουσία. Κάτι άλλο που βλέπουμε, να αλλάζει δηλαδή η αντίληψη του κοινού, είναι συντονισμένες επιθέσεις hackers σε οικονομικούς θεσμούς, σε τρεις βαλκανικές χώρες, που δείχνουν ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις ε, επιθέσεις αυτές και επομένως δημιουργούν ένα περιφερειακό οργανισμό με ένα κοινό κέντρο για την αντιμετώπιση επιθέσεων hacker. Εν τέλει, πάντα σύμφωνα με το σενάριο, καθώς συνεχίζει η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένταξη, γίνονται μεταρρυθμίσεις και πραγματικές μεταρρυθμίσεις και φτάνουμε στο σημείο 2025, όπου το Μαυροβούριο εντάσσεται, γίνονται ορταστικές εκδηλώσεις στην Ποντγκόριτσα κλπ και οι υπόλοιπε χώρε θεωρούν ότι έχουν καθαρό, καθαρή ε, ε, μονοπάτι μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο σενάριο τώρα. Παρέμβαση της σερβικής intelligence σε γειτονικέ χώρε. στοιχεία του βαθέως κράτους που, είναι, ε, που υπάρχουν μέσα και στις υπηρεσίες αυτές και που δεν έχουν μεταρρυθμιστεί και που είναι απολύτως φιλορωσικά υποστήριξη της ε, Μόσχας σε οποιαδήποτε πολιτική που παρεκκλίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ανταμοιβή μάλιστα από τη Ρωσία οικονομική υποστήριξη για τους ακροδεξιού οργανισμούς, αυξημένος μάλιστα, αλλά περιορισμένη οικονομική επιρροή. Διότι η Ρωσία δεν μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα από οικονομική άποψη. Η ήπια δύναμη σε υπερβολικό βαθμό λόγω εθνικών ε, διαφορών, ε, αυτή είναι η μεσαία περίπτωση. Το 2025 δηλαδή ε, οι περισσότερες χώρες δεν θα είναι πολύ κοντά στο να γίνουν μέλη και περισσότερο κατάσταση θα έχει μείνει με, ίδια με τη σημερινή. Αλλά αυτό που είναι σημερινό για αυτό, ε, σημαντικό για αυτό το σενάριο και τη ρωσική επιρροή είναι ότι και αυτό το σενάριο είναι η χειρότερη περίπτωση, διότι το status quo μπορεί να διατηρηθεί μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι ότου εκραγεί και εξελιχθεί σε κάτι πιο επικίνδυνο. Και πάμε τελικά στο χειρότερο σενάριο που φαίνεται να τραβάει και τη μεγαλύτερη προσοχή εδώ θα έχουμε ένα Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών παρόντα σε στρατιωτική παρέλαση στην Πανιαλούκα ε, για τον εορτασμό της ανεξαρτησίας της Ρεπουμπλικας Εύσκα. Πώς στάσαμε εκεί, ξεκινώντας με διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Η Σερβία υπόσχεται ότι θα ζητήσει από τη Ρωσία να μην μπλοκάρει το, να γίνει το κοσυφό πεδίο μέλος του ΝΑΤΟ. Σχεδιάζονται και καθιερώνονται σύνορα. Η στιγμή της αλήθειας φτάνει το κοσυφό Κάνει αίτηση για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απορρίπτεται και η Ρωσία λέει ότι δεν μπορεί να δεχθεί να είναι το κοσυφό μέλο μέλος των ΗΠΑ. Αυτό εντείνει την κατάσταση στη Σερβία και στο Κωσυφοπαίδιο και η ακροδεξιά στη Σερβία ανεβαίνει διότι λέει ότι η χώρα έχει πουληθεί σε προδότες, ότι όλη η συμφωνία με το Κωσυφοπέδιο δεν χρειαζόταν να γίνει. Στο Κωσυφοπέδιο υπάρχει κρίση διακυβέρνησης και απώλεια ε, εδαφών αυξάνεται η με τη Ρωσία. Η Ρωσία παρέχει τώρα σήμερα ένα πλαίσιο ασφαλείας μαζί με την Τουρκία στις χώρες αυτές και η Ευρώπη και να σας δώσω μια παράθεση από το κέρμα αυτό, κάτι που λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ανώτατο Συμβούλιο το 2024 επισκεπτόμενος για πρώτη φορά την, την Πανιαλούκα για την πρώτη επέτειο ανεξαρτησίας λέει η Ευρώπη απέτυχε ξανά να φέρει την έρευνα στα Βαλκάνια. Ορισμένοι ερωτιούνται κατά πόσο το έχει κάνει επίτηδε. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς κάποιο τέτοιο σενάριο σε τελική ανάλυση, σε αυτό το σενάριο όπω και στα υπόλοιπα που μπορείτε να διαβάσετε στην έκθεση. Υπάρχει αλλαγή κυβέρνηση στο Μαυροβούνιο με μια πρόρωσική κυβέρνηση στα Ηνία, ε, μια προσπάθεια επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό λόγω τη ε, απόπειρα συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και αποτυχία επίτευξη συμφωνία τελικά πρόρωσική κυβέρνηση στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στη Σερβία και έτσι υπάρχουν τρει χώρες στα Βαλκάνια με προ-ρωσική στάση και φυσικά σε, πολύ μακριά από το να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπερασματικά αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε φορά που η Ευρώπη ε, δεν ε, κάνει κάτι γεμίζει το κενό η Ρωσία. Παίζει κάποιο σταθεροποιητικό ρόλο αφενός, αφετέρου όμως δεν υπάρχει καμία αναλλακτική σε σχέση με αυτά που προσφέρει η Ρωσία. Εξακολουθεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλή θέση στην περιοχή και αυτή θα πρέπει να την παγιώσουμε. Τι είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που ακούσαμε ήδη εδώ, όχι να εστιαστούμε απαραίτητα στην ίδια τη Ρωσία μόνο, αλλά και στα προβλήματα, στις ταραχές που δημιουργούν προβλήματα στις χώρες αυτές και ανοίγουν το δρόμο για τις ε, ε, για τη Ρωσία, επίλυση διμερών ζητημάτων, ζητήματα ασφαλείας, ενίσχυση της διακυβέρνησης του κράτους δικαίου που αλλιώς ανοίγει τους δρόμου για την Κίνα, για τη Ρωσία να ασκήσουν επιρροή που δεν θα μπορούσαν να είχαν ασκήσει διαφορετικά αν δεν υπήρχαν τέτοια κενά σε αυτούς του τομεί. Ενίσχυση της οικονομικής ε, ε, μετάβαση και βελτίωσης. Ε, έχω και μία ιστορία από την EAS. Δημοσίευσαν ένα βιβλίο για παιδιά για τον πολιτισμό, πολύ καλά σχεδιασμένο που εξηγεί πόσο κοντά βρίσκονται η Ευρώπη με τα Βαλκάνια. Και αυτό εμένα με ενθουσίασε. Πώς δηλαδή με δημιουργικούς τρόπους μπορούμε να σχεδιάσουμε τη συνεργασία και την επικοινωνία. Και τέλος το να είμαστε παρόντες. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να πάει ποτέ να είναι παρούσα και να είναι ο ισχυρότερος φορέας, ισχυρότερος παίκτη στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεπέρκοβιτς για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ε, και θα μοιράσουμε την ε, έκθεσή σας στα μέλη αν ε, συμφωνείτε τώρα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ, Κλέρ, και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και εγώ τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες αγωγικές τους παρατηρήσεις και ίσως θα ήταν καλό να ακολουθήσει Ακολουθήσω κάποιε ερωτήσει και απαντήσει. Καταρχήν, θα ήθελα να κάνω την εξή παρατήρηση. Εδώ και τέσσερα χρόνια παρακολουθώ τι εξελίξει στην περιοχή τη Βαλκανική. Ω ε, ε, εισηγητή στι ε, διαπραγματεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σερβία. Και έχω τέσσερι ερωτήσει. Η πρώτη είναι η εξή. Ευσταθεί η εντύπωσή μου ότι προφανώς ε, το, η προσπάθεια πραξικοπήματος εκ μέρους της ε, Ρωσίας στο Μαυροβούνιο δεν έτυχε κάποια επαρκούς αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι απίστευτο ε, ένα κυρίαρχο κράτος, σε ένα κυρίαρχο κράτος γίνεται προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης εκ μέρους της Ρωσίας. Ποια είναι η δική σας εντύπωση, γιατί έγινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ε, έγινε πολύ λόγος για το ρόλο του κυρίου Ντόντικ στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Πολύ συχνά έχουμε συζητήσει για το ρόλο που παίζει ο κύριος Ντόντικ στη χώρα αυτή και συχνά συζητούμε τι είδου ε, απειλή ε, συνιστά για την ενότητα της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Από την άλλη, πώς αντιμετωπίζετε τις πρόσφατες εξελίξεις ότι οι Κροάτες στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ε, έχουν ε, συμμαχίσει με τον κύριο Ντόντιτς. Ε, και ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν, προσπαθούν να σπρώξουν τους Κροάτες στις αγκάλες του κυρίου Ντόντιτς. Γιατί οι Κροάτες ε, είναι ξανά συνδεμένοι με, τα, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ε, τρίτον, ε, γίνεται πολύ λόγος για την επιτυχία του Σπούτνικ. Εμείς προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τις δικές μας δραστηριότητες, για παράδειγμα του BBC, της Deutsche Welle. Ε, τι παρατηρείτε σε αυτή τη στιγμή, έχουν αυξήσει την επιρροή τους, έχει, έχουν αυξήσει τα ποστά της ακροματικότητας και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε προκειμένου να αντισταθμίσουμε τη ρώσικη προπαγάνδα μέσω του Sputnik. Επίσης, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσει ε, ε, μια δημοσιογραφία υψηλή ποιότητας στα Δυτικά Βαλκάνια. Πώς θα μπορούσαμε ε, να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τους σπουδάζοντες, τους επαγγελματίες δημοσιογραφίες στις χώρες αυτές προκειμένου να προσπαθήσουν να είναι πιο αμερόληπτοι. Okay. Uh, there's a fairly comprehensive set of questions. Πολύ καλές ερωτήσεις. Ε, αν θέλετε να ξεκινήσετε, έχετε εξή μια ερώτηση. Ναι, κάποιες από τις ε, ερωτήσεις που είχαμε στο μυαλό μα, τις έκανε και ο Ντέβιτ Μακαλιστερίδη. Ήθελα να προσθέσω άλλη μία. Είπατε ότι η Ρωσία δραστηριοποιείται σε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δραστηριοποιείται παρκώς στην περιοχή. Ωστόσο, τα κράτη στα Δυτικά Βαλκάνια δεν παρουσιάζουν και αυτά ορισμένα ελλείμματα όσον αφορά την ανάπτυξη της κοινωνίας και της πολιτικής. Και εκεί δεν υπάρχουν κάποια κενά που αποτελούν πρόσκληση για κάποια ξένη επιρροή. Ευχαριστούμε, Ρεμπέκα. Κύριε Τσάρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για, ε, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τις παρουσιάσεις σας και για τα όσα είπατε για τη ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια. Έχω ένα γενικό σχόλιο και θα ήθελα να αντιδράσετε σε αυτό που θα πω. Η Ρωσία πράγματι ασκεί την πολιτική της και κάποιος είπε ότι πρόκειται για έναν χονδροειδή συντηρητισμό. Η Ρωσία συχνά παρουσιάζεται ως υπερασπιστής των χριστιανικών αξιών και πολύ συχνά πίσω από αυτό βρίσκονται πρώην αξιωματούχοι του KGB και χρησιμοποιούν τη γλώσσα του Λένιν προσπαθώντας να βρουν τα αδύναμα σημεία, τα τροτά σημεία των ε, εχθρών. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις, δεν πάβει να είναι γεγονό ότι χρησιμοποιούν την προπαγάνδα αυτή κατά οποιοδήποτε αντιτίθεση στις χριστιανικές αξίες. Ξέρουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις θρησκείες, οπότε δεν κάνει εντύπωση που η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά των φιλελεύθερων τάσεων. Αυτή είναι η τάση της Ορθόδοξης του Ορθόδοξου Χριστιανισμού είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση. Η Ρουμανία τώρα που είναι ένας από τους μεγαλύτερους γείτονες της Σερβίας όταν ακούμε για το ομοφοβικό δημοψήφισμα στη Ρουμανία και μετά το συγκρίνουμε με την δραστηριοποίηση των Ευρωπαίων ε, επιτρόπων και τις δραστηριότητε τους πριν από το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Όλα αυτά είναι επιχειρήματα που βοηθούν τη ρωσική προπαγάνδα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να πείσουμε τους συνανθρώπους, τους συνανθρώπους μας στα Δυτικά Βαλκάνια απλά πρέπει να απέχουμε από τέτοιες δραστηριότητες να εγκαταλείψουμε τι δραστηριότητες αυτές γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιχειρήματα που στηρίζουν τη ρωσική προπαγάνδα κατά του δυτικού κόσμου. Κάτι που αποτελεί γεγονός. Εγώ έχω ήδη απευθύνει έκκληση για επικοδομητικό διάλογο με τις εκκλησίες στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με τους θρησκευτικού εκπροσώπους. Πρέπει τις θρησκείες να τις αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ως θεσμούς, αλλά και να τους προσφέρουμε και κάτι. Αυτές ήταν και ο φορέας που βοήθησε στην αντίθεση του λαού κατά του κομμουνισμού. Στις δυτικές χώρες έχουμε φυσικά την πολυμορφία των αξιών και κάποιοι πολιτικοί διαφορετικών απόψεων μπορεί να μην το υποστηρίξουν αυτό, αλλά εδώ έχουμε πολλούς συντηρητικούς και ο συντηρητισμός αφορά ουσιαστικά το σεβασμό κάποιων αξιών. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν και να αντιδράσουμε σε αυτή τη χοντροειδή προπαγάνδα της ρωσικής πλευράς. η δική μας πίστη του δικού μας πολιτισμού, προς το δικό μας πολιτισμό είναι το καλύτερο επιχείρημα που έχουμε για να πείσουμε τους ανθρώπους που ανέκαθεν υποστήριζαν το δυτικό πολιτισμό. Ευχαριστώ. Thank you. And now, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Σκόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να προσθέσω και κάτι σε αυτά που είπαν η Ρεμπέκα και ο Ντέιβιντ. Η προπαγάνδα, αυτή η προσέγγιση των Ρώσων είναι πολύ εκλεπτισμένη και στρέφεται κατά όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πολύ στοχευμένη η προσέγγιση. Ψάχνουν να βρουν τα πιο ευαίσθητα θέματα σε κάθε χώρα και στοχεύουν ακριβώς αυτά. Θρησκεία, μετανάστευση, κοινωνικά ζητήματα. Ευαίσθητα θέματα για τους πολίτες και τι λένε, κοιτάξτε, το κακό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν ανήκετε σε αυτούς. Τους λένε, ανήκετε στον πραγματικό χριστιανισμό. Την όλη ιστορία την ξέρουμε και είναι εύκολο και ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς πώς άλλαξαν, να μετασχημάτισαν ουσιαστικά την ιδεολογία του λεμινισμού, του μαρξισμού σε ε, κάτι που υποστηρίζει την τον ορθόδοξο χριστιανισμό της Μόσχας. Ποια είναι η συνταγή? Τι να κάνουμε εμείς ως Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκρούσουμε αυτή την πολύ πραγματικά εκλεπτισμένη προπαγάνδα κατά των χωρών μας. Ξέρουμε ότι και μάλιστα είχαμε ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο για την επιρροή των τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δυστυχώ η αριστερά και δεν βλέπω να είναι κανεί εδώ από του σοσιαλιστέ, και αυτό είναι και καλό σημάδι. Μόνο εσεί. Η ομάδα σα δεν είναι και απήχε κατά τη διαρκή της ψηφοφορίας για το ψήφισμα αυτό. Υπήρχαν και διάφορε ψευδεί ειδήσει σε σχέση με αυτό το ψήφισμα. Κατηγορήθηκα ότι ψήφισα κατά του χριστιανισμού και διάφορα τέτοια. Αλλά εδώ πρέπει να δείξουμε ε, ε, ότι είμαστε ενωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί του θέματος αυτού. Είναι απολύτως αναγκαίο, θεωρώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συμβάλλω στη ζήτηση αυτή. Είχατε λεπτομερείς ε, ερωτήσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσετε. Αλλά τονίζοντας ε, τα όσα είπε ο Ντέιβιτ, Εν σχέση με την ε, ε, εκπαίδευση νέων δημοσιογράφων ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον, να υποστηρίξουμε την ποιοτική δημοσιογραφία. Αλλά θα θέλαμε να μας πείτε τη δική σας αξιολόγηση για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επικοινωνίες προς τους πολίτες της χώρες αυτές. Πόσο αποτελεσματικοί έχουμε υπάρξει και τι τι περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση στο πεδίο αυτό. Ε, θα ακολουθήσει τη σειρά που μιλήσατε αρχικά. Ε, πολλές ερωτήσεις μου απευθύνεται. Δεν θα απαντήσω σε όλες. Γιατί το αποτυχημένο τι έγινε με το αποτυχημένο πραξικόπημα στο Μαυροβούνιο. Νομίζω ότι φταίνε οι αρχές του Μαυροβουνίου γιατί ε, ε, έγινε ένα πραξικόπημα για πολιτικές σκοπιμότητες. Σήμερα έχουμε έναν άλλον επικεφαλής αντιπολίτευσης ο οποίος συνελήφθη. Παρακαλώ μην με παρανοήσετε. Εγώ, εάν ήμουν Μαυροβούνιος, δεν θα ψήφισα ποτέ την αντιπολίτευση. Αλλά όταν ε, κανείς ε, στραγγαλεί στους πολιτικούς του αντιπάλους, δημιουργεί το πεδίο παρέμβασης των ε, Ρώσων. Αναμέναμε ενδιαφέρον τα συμπεράσματα ε, της εισαγγελία ε, για το πραξικόπημα στο Μαυροβούνιο, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό διαπαντός. Ε, ως, ε, αυτό και για να αυξηθεί η αποξεπιστία του Μαυροβουνίου, αλλά και για να ενισχυθεί η δημοκρατία εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι στο Μοντενέγκρο δεν υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Στη Βοσνία η Ρωσία ε, παίζει πολύ ενδιαφέρον ε, παιχνίδι. Ε, σκεφτόμαστε τους κράτες ως εχθρούς της Ρωσίας. Αλλά η Ρωσία δεν έχει φίλους και εχθρούς, έχει τέρους. και μπορεί αύριο να σφυλατήσει μια συμμαχία με κάποιον που δεν τον περιμένει κανείς. Ε, και ε, διάφοροι Κροάτες έχουν αμβλύνει τη ρητορία τους ε, εναντίον της Ρωσία, απέναντι στη Ρωσία. Η Ρωσία, κατά την άποψή μου, δεν έχει καμία ιδεολογία. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πρόθεση των, των συμφερόντων της. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, λέτε, να ενισχύσει την ε, υψηλή ποιότητα δημοσιογραφίας. Ε, και μάλιστα χώρε μέλη, γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα εργαλεία. Ε, την, όταν ο κύριος Βούτσιτς τολμά να προκαλέσει τις αρχές, κανείς ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτές τις αξίες και τις αρχές. Ε, γιατί έγινε αναφορά στις ε, ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Έχουν μεν τη δημοκρατική νομιμότητα οι θύνοντες εκεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο οι δημοκρατικές αρχές. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ε, πληρώνει για τα ΜΜΕ και λοιπά. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να μπορούμε να χρηματίσουμε τον, τη ροή των ε, χρημάτων. Στην ε, ε Σερβία συνήθως υπάρχουν ταυτόσιμα πρωτοσέλιδα. Ναι, θα πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση των νέων δημοσιογράφων προκειμένου να καλλιεργήσουν τις αξίες τις οποίες υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Ε, Υπάρχει μια παρουσία των δυτικών με μια ε, το CNN για παράδειγμα, λειτουργεί τοπικά. Ε, και μπορεί κανείς βεβαίως να πει ότι έκαναν μεγαλύτερη επένδυση από τους ε, Ρώσους. Τώρα θα πω κάτι για την Τουρκία Ορισμένοι δημοσιογράφοι ταυτίζουν, βάζουν το ίδιο καλά τη Ρωσία με την Τουρκία, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία έχει ένα πολύ αμφίσιμο ρόλο. Βεβαίως ε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θέλει να έχει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, αλλά είναι και στο ΝΑΤΟ, αλλά και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση. Εάν ε, το δούμε μακροπρόθεσμα, η Τουρκία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στο ίδιο οικονομικό μπλοκ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν συμμερίζεται ίσως τις ίδιες αξίες, αλλά ανήκει στο ίδιο μπλοκ. Ενώ η Ρωσία όχι. Ε, και τα, όταν ο κύριος... Ε, who have their cousins, ε, Όταν πάει ο Ερντογκάν στο Σιντζάκ, τον συναντούν χιλιάδες. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, υπάρχουν πολλές ε, συλλογικότητες ε. και υπάρχει και ένας κοινό παρανομαστής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι διαφορετική η περίπτωση Τουρκίας από τη Ρωσία. Δεν ταυτίζονται. Εγώ, θα πήγαινα, θα πάω ανάποδα μάλλον, θα αφήσω το Μαυροβούνιο για το τέλος. Πρώτα, ρόλος της Ρωσίας στην Βαλκανική. Μπορεί να μην είναι τίποτα το νέο αυτό που θα πω, αλλά ε, υπενθυμίζοντας το όσα είπαν οι συναδελφοί μου, παίζει το ρόλο spoiler, δηλαδή ψάχνει να βρει τα κενά για να βάλει σφήνε ανάμεσα στις χώρες. Δηλαδή θα υποστήριξει την Σερβία κατά της Αλβανίας στο Κόσοβο, τα Βόσνιους ε, Είναι λοιπόν η ιδιώδης κατάσταση που για τη Ρωσία θα ήταν ε, να υπάρξει άλλη μια κατάσταση ε, παγωμένων συγκρούσεων. Διότι όσο υπάρχει αυτό που είναι πραγματικά πρωταθλητής η Ρωσία και όσο το περισσότερο κρατούν τόσο καλύτερα. Αντίθετα λοιπόν με την Κίνα που παίζει διαφορετικό παιχνίδι, η Κίνα εποφελείται από την διαδικασία διεύρυνσης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα θέλει σταθερά περιβάλλοντα για να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Που τελικώς πάνε να πέσουν στην παγίδα οι περιοχές αυτές. Για παράδειγμα, 2 δισεκατομμύρια στην Σερβία, ε, στο Μαυροπόνιο λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο. Όμως η Κίνα δεν καταστρέφει, εμφανίζεται ως μια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή, διότι διαθέτει χρήματα που χρειάζονται οι χώρες της Βαλκανικής. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, θρησκεία και τις σχετικές αξίες, ο Μακεβέλη είπε κάποτε, αν δεν μπορείς να πετύχεις με άλλο τρόπο, Στρέψω στη θρησκεία. Εγώ συμφωνώ ότι η θρησκεία και η πολιτική πάνε χέρι με χέρι μια χαρά μαζί και γνωρίζω ότι συχνά είναι η Ρωσία πίσω από το αφήγημα αξιωματούχοι της ΚΑΓΚΕΜΠΕ οι οποίοι ποτέ δεν υπήρξαν θρήσκοι και ακόμη και σήμερα η πίστη του στη θρησκεία είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμη. Θυμίζω όμω ένα πράγμα. Υπάρχει μια θρησκευτική επιτροπή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας που συναποτελείται από μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αξιωματούχους και που συνεργάζονται πολύ στενά για να αυξήσουν την επιρροή της Ρωσίας στον Ορθόδοξο, κόσμο. Έτσι χρησιμοποιεί η Ρωσία την θρησκεία για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και έρχομαι στο ερώτημα της εκπαίδευσης, παιδείας. Η παιδεία ως μηχανισμός, όχι μόνο δηλαδή να εκπαιδεύσουν ανθρώπους, ας πούμε, ανθρώπους, δημοσιογράφους για παράδειγμα, για να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι ψευδείς πληροφορίες κλπ, ποιες είναι φτιαγμένες πληροφορίες, ειδήσει, αλλά να εκπαιδευτούν και σχετικά με τις αξίες, τις αξίες του δυτικού κόσμου. Γιατί είναι σημαντικό για μας να βρεθούμε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ανταγωνιστεί επιτυχώς με Ρωσία και Κίνα και άλλους θα πρέπει να αλλάξει λίγο το αφήγημα και να δώσει περισσότερη έμφαση στο συνέστημα, διότι τι κάνει η Κίνα. Με χρήματα, διότι όλες οι χώρες αυτές δέχονται δάνεια από την Κίνα. Όχι όμως άμεσες επενδύσεις, δάνεια που δίνονται σε κινέζικες εταιρείες για έργα κατασκευών στην Βαλκανική. Και από αυτά τα χρήματα οι Κινέζοι τι κάνουν, φτιάχνουν, ας πούμε, εξοπλίζουν ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο, εμφανιζόμενοι έτσι σαν κάποιοι οι οποίοι βοηθούν του απλούς ανθρώπους και αυτό λειτουργεί μια χαρά. Προσπαθώ τώρα ε, να ερευνήσω εδώ και μήνες τον ρόλο της Κίνας στη Βαλκανική και πιστέψτε μου δεν βρήκα ούτε ένα άρθρο αρνητικό σε Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σερβία κλπ αρνητικό για τους Κινέζους. Για όλους, όλα τα νέα, όλες οι ειδήσει δείχνουν ότι οι Κινέζοι είναι φιλικοί, θετικοί και βοηθούν. Τώρα, για το Μαυροβούνιο. Θέμα περίπλοκο. Και συμφωνώ. Κάτι που καθιστά δύσκολο για ορισμένε χώρε να αντιληφθούν περί τίνο πρόκειται. Έκανα μια σχετική έρευνα και έχω γράψει και μια έκθεση για το ΝΑΤΟ το 2016. Και εγώ στην αρχή πίστεψα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Σαν τους παγίδευσαν. Αλλά πρέπει να πω τώρα μας βοήθησε πολύ η υπηρεσία πληροφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αξιωματούχοι της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και για τη δικαστική διαδικασία που είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για πολλούς λόγους και για τη δημοκρατική διαδικασία στο Μαυροβούνιο και για την δημιουργία θεσμών και ελπίζω ότι τελικώς θα φωτιστεί η υπόθεση. Όμως όσο διαφεύγουν αυτοί οι δύο είναι δύσκολο να κλείσει η υπόθεση. Ευχαριστώ κύριε Σεβέρκοβιτς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν για τον Ντόντιτς και τους Κροάτες στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Τα έχουμε αυτά και στο ένα από τα σενάριά μας. Ότι δηλαδή συνεργάζονται αυτοί οι δύο για να διαλυθεί εντελώς η Βοσνία Ζεγοβίνη. Και κάτι το οποίο ε, έχει λογική. Αν προσπαθήσει κανείς να διαλύσει μια χώρα και σε αυτή συναπαρτίζεται από τρία μέρη, τότε δύο αρκούν να συνεργαστούν για να διαλυθεί. Για τη δημοσιογραφία. Μπορεί να πει κανεί ότι είναι καλό να έχουμε καλά προγράμματα για να ενθαρρύνουμε ε, και να βελτιώσουμε την ενημέρωση των δημοσιογράφων, πώς να γράφουν πιο σωστά τις ειδήσει και πιο αληθινές. Και ε, υπάρχει και ο ρόλος της δημοσιογραφίας στην ανάπτυξη, ανάδειξη ορισμένων πολιτικών κομμάτων, αλλά αυτό που φάνηκε είναι ότι οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν και δύο άλλα θέματα τα οποία κρύβονται εκεί, δηλαδή η λογοκρισία soft ή ε, ισχυρή ή αυστηρή και υπάρχουν και σπάνια στοιχεία σκληρής λογοκρισίας δηλαδή δεν είναι κάπου ένας λογοκριτής που να λέει στο γραφείο ότι αυτό δεν μπορεί να δημοσιευτεί οι συντάκτες γνωρίζουν τι μπορεί να δημοσιευτεί και τι όχι επομένως δεν χρειάζεται να εμπλακεί κανένας και πώς το γνωρίζουν αυτό διότι όπως είπε και ο Ντίμηταρ ακολουθούν το χρήμα ξέρουν όπου προέρχεται το χρήμα και σύμφωνα με το κριτήριο αυτό λαμβάνουν κάποιε αποφάσεις. Στη Σερβία ένας από τους ηγέτε της αντιπολίτευσης δέχθηκε επίθεση πριν από λίγε ημέρες και χρειάστηκε μια ολόκληρη ημέρα το κεντρικό δημοσιογραφικό ε, όργανο να πει κάτι γι' αυτό. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να το δει κανεί ή ότι οι δημοσιογράφοι δεν το γνωρίζουν. Αυτό που θα προτείνω εγώ είναι η τη της στήριξης προγραμμάτων υπέρ των δημοσιογράφων και βέβαια ε, επενδύσεις στην καλή δημοσιογραφία και υπάρχουν, υπάρχουν τέτοια, υπάρχει και πλήθος ε, ανθρώπων που λειτουργούν πάρα πολύ καλά, έστω και με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, πρέπει ωστόσο να ρηχτεί βάρος στην εκπαίδευση της νεότερης γενιάς και να αντιλαμβάνονται και οι αναγνώστες τι συμβαίνει. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Και αυτό με φέρνει σε ένα τελευταίο θέμα. Τα Βαλκάνια δεν είναι καμία ειδική περίπτωση. Είναι μια περιοχή η οποία περνά μέσα από μια μεταβατική περίοδο, η οποία δεν έχει λήξει και ε, μια ε, περιοχή η οποία κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της μεταβατικής περίοδου της. Και ε, η αναζήτησή μας είναι ποιο θα είναι η τελική έκβαση αυτής της μεταβατικής περίοδου. Και αυτό είναι, αυτά είναι τα σενάρια μας για το 2025. Τέλος, για την παρουσία άλλων παραγόντων, όχι αναγκαία των Ρώσων. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε για την Τουρκία και την τουρκική επιρροή, ότι ως τώρα δεν έχουμε δει αρνητική επιρροή των Τούρκων στα Βαλκάνια. Θα αλλάξει αυτό, γιατί δεν το ξέρουμε. Αρνητική επιρροή λέτε κύριε Μακάλιστερ. Καλά, σύμφωνοι, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εννοούσα σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής ένταξης και πώς αντιμετωπίζουν τις πτυχές αυτής, όχι, όχι για θέματα ε, κοινωνίας. Κοινωνία, βεβαίως. Ε, ε, συγγνώμη, Κίνα, πώς το λένε, Κίνα, Κίνα. Πάρα πολύ ε, σημαντικός οικονομικός παράγοντας. Και η Ρωσία είναι ιδιαίτερη περίπτωση ό,τι αφορά τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί. Τέλος. πότε είναι υπερβολικά δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε ενδεχομένω θα υποχωρήσει και τι μπορεί να γίνει στο προσεχέ μέλλον. Μία περίπτωση μπορεί να είναι η κατάσταση μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου και πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση. Εκεί θα είναι σημαντική στιγμή για να επανέλθει η Ρωσία στο πλαίσιο των Βαλκανίων και καθοριστική στιγμή, κατά τη γνώμη μου, για το πώ θα προχωρήσουμε σχετικά με το τι σημαίνει η Ρωσία για την Σερβία και τι σημαίνει η Ρωσία για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Αν δεν έχετε κάποια άλλα σχόλια ή κάποιες παρατηρήσεις, ε, θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη και των δύο επιτροπών μας για τη συμβολή σας. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πολύ διαφωτιστική για μια κατάσταση σε ταχεία εξέλιξη, ε, όπου απομένουν να γίνουν πολλά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ξανά και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Στην παρούσα λοιπόν ε, κλείνουμε την ακρόαση αυτή. Mm να ρωτήσω τους συναδέλφους, υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε από τα διάφορα. Όχι, από όσο ξέρω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και κλείνουμε την σημερινή συνεδρίαση.